Diamo inizio al nostro workshop. Θα ήθελα να ξεκινήσει παρακαλώ το εργαστήριο μελέτης. Παρακαλώ καθίστε. Innanzitutto voglio ringraziare Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους ε, παρευρισκόμενους του τους εκπροσώπους ε, των ε, οργανώσεων, αυτούς που διοργάνωσαν ε, την, το εργαστήρι, τους εισηγητές που θα παρέμβουν σήμερα. Ευχαριστώ ιδιαίτερο τη Μαριάν Φίσερ Μπολ, τον Έσκιλ Άντερσον, Υπουργό της Σουηδίας για θέματα γεωργίας που δέχτηκε αυτή την ε, πρόσκληση. Αυτό το σεμινάριο μας δίνει την ευκαιρία να ανοίξουμε μια, ένα ουσιαστικό παράθυρο για να εμβαθύνουμε το, για το μέλλον της, πολιτικής, ε, της γεωργικής πολιτικής. Το κάνουμε μια δύσκολη στιγμή ε, που συμπίπτει με τον προβληματισμό για τον κοινοτικό προπολογισμό και που δυστυχώς εκθέτει την ΚΑΠ σε κίνδυνο μειωμένων κονδυλίων καταρχάς ε, ανταγωνισμό από άλλες πολιτικές ε, που διεκδικούν και αυτές προπολογισμό και από την άλλη τις πρώτες θέσεις που, έχουν, που έχει πάρει πάνω στο θέμα αυτό η Κομισιόν ότι και αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να ε, λάβουν άλλου, άλλης διάστασης κονδύλια. Σήμερα είναι η μόνη οικονομική πολιτική, η γεωργική δηλαδή, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, που είναι πραγματικά κοινο, κοινοτική. Ε, και είναι η πιο σημαντική πολιτική διαχείριση των εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε στην, στο κλείσιμο της διαδικασίας επικύρωσης της Συνθήκης Λισαβόνας και αυτή είναι μια ιστορική στιγμή στις διαθεσμικές σχέσεις δίνει περισσότερη εξουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα γίνει επιτέλους ε, αποφασιστικός εταίρος στην ε, διαδικασία παραγωγής νομοθετημάτων και για γεωργικά θέματα. Ε, σήμερα έχουμε αυτή την ευκαιρία ε, να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα και ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί θα παίξουμε ε, ένα ρόλο πάρα πολύ σημαντικό και εκ των κάνευ στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Πρέπει να δούμε το μέλλον της γεωργικής πολιτικής. Καθώς εξελίσσεται η ΚΑΠ, ε, μπαίνουν καινούργια θέματα ε, που οφείλονται στις αλλαγές της κοινωνία μας. Νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία, οι θεσμοί της και οι πολιτικές της. Η πολιτική για τα γεωργικά θέματα είναι ε, βασικός παράγοντας ε, της ε, οικοδόμησης της Ευρώπης και σήμερα ο ρόλος της, οικονομικός και ρόλος διαχείρισης των εδαφών είναι πολύ πιο σημαντικός. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση στις νέες παγκόσμιες προκλήσεις, πισιτιστική ασφάλεια και βιωσιμότητα των διαδικασιών ανάπτυξης πάνω απ' όλα θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στη γεωργική πολιτική για να μειωθούν ε, οι όποιες τρευλώσεις. Υπάρχει ανάγκη να αντιμετωπίσουμε νέες παγκόσμιες ευθύνες και πραγματικά η γεωργία μπορεί να παίξει εκεί ένα σημαντικό ρόλο. Μία επιτάχυση της διαδικασίας μεταρρύθμισης της ΚΑΠ έχει ε, ήδη προβλεφθεί ε, στη μεταρρύθμιση του 2003 και με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να μειωθούν η προστασία, θα πρέπει να μειωθεί η προστασία των αγορών ε, και να προωθηθεί η στήριξη των τιμών. Θα πρέπει η πρημοδότηση προς τον Γεωργό να αντικατασταθεί από μια πρημοδότηση με βάση τη συμπεριφορά και τις υπηρεσίες που προσφέρει στην κοινωνία. Αυτή η νέα φιλοσοφία είναι πάρα πολύ επίκαιρη μετά από τις ε, αλλαγές που έχουν ε, βάλει το αποτύπωμά τους ε, στις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων. Όμως, αυτές οι νέες προκλήσεις μπορεί να υποσκάψουν την αγροτική πολιτική θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη συζήτηση που, γίνεται για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, όπως προκύπτει από το non-paper της Κομισιόν. Ε, νομίζω ότι αυτό το κείμενο δεν πηγαίνει προς την ε, σωστή κατεύθυνση. Είναι άτυπο κείμενο και επομένως δεν εκδηλώνει τη βούληση της Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά το περιεχόμενο ε, συζητήθηκε ευρέως. Οι ίδιες ε, επιλογές ε, του να συζητήσουμε δηλαδή τον προπολογισμό πριν συζητήσουμε την ίδια την αγροτική πολιτική δεν είναι σωστό. Να, το να προτάξουμε τη λογιστική πέρα και πριν από, τα, από το περιεχόμενο δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Γιατί ζούμε μια ιστορική στιγμή στις κοινωνίες μας. Η ανάλυση που γίνεται στο σχέδιο ανακοίνωση ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση και εκμοντερνισμό των γεωργικών δαπανών ε, μοιάζει να έχει αντιφάσει σε πολλά σημεία και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η αξιολόγηση που θα μας κάνει η Επίτροπος. Θα πρέπει να δούμε πώς θα ενδυναμώσουμε το περιεχόμενο της ε, γεωργίας, πώς θα τη βοηθήσουμε ε, για να μας βοηθήσει στον αγώνα κατά των αλλαγών του κλίματος, ε, στον αγώνα αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στο να προωθήσουμε τις ε, προσδοκίες της κοινωνίας, ε, τη βιοπικιλότητα, την ευμερία των ζώων και την χρήση των υδάτινων πόρων. Φυσικά, ταυτόχρονα φαίνεται περίεργο που σε αυτό το κείμενο γίνεται σαφής αναφορά σε μια μεγαλύτερη ευθύνη των κρατών μελών στο εσωτερικό του... για τα θέματα δαπανών για τις ε, ΚΑΠ. Και επομένως είναι σε αντίφαση με τις ε, θέσεις του Κοινοβουλίου που λέει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επαναπατρισμού εντός εισαγωγικών της ΠΑΚ ό,τι αφορά την εισαγωγή της ε, συγχρηματοδότησης στον πρώτο πυλώνα της στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα της ΚΑΠ θα δημιουργήσει μεγάλες ανισορροπίες ε, στον γεωργικό τομέα και σε αυτή τη φάση της ε, κρίσης τα πιο φτωχά κράτη-μέλη θα έχουν δυσκολίες για να χρηματοδοτήσουν ε, την γεωργία. Δεν θέλω να κάνω βέβαια μια ανάλυση του εγγράφου, αλλά θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν φοβεροί κίνδυνοι που συνδέονται με αυτές τις ε, κατευθύνσεις του κειμένου. Επιμένως, ε, από την άλλη, η κρίση στον ε, γαλακτοκομικό τομέα δείχνει ότι το να μειώσουμε τις, τα έξοδα, για την, τις δαπάνες για την ΚΑΠ δεν σημαίνει ότι θα ξοδεύουμε λιγότερο στην Ευρώπη για τη γεωργία, αλλά αντίθετα θα, θα αυξήσουμε τους, τα κονδύλια τα οποία επενδύουμε τα οποία δεν δίνουν αποτελέσματα. Και επιπλέον θα υπάρξουν και φοβερές ανισορροπίες στη μεταχείριση των γεωργών. Κλείνω λέγοντας ότι έχουμε μια θεώρηση εντελώς δημοσιονομική. Ε, νομίζω ότι η θέση της Κομισιόν θα μπορούσε να επανισορροπηθεί λαμβάνοντας υπόψη την δουλειά του Κοινοβουλίου. Η θέση σε ισχύ της Λισαβόνας από 1η Δεκεμβρίου του 2009 δείχνει, ε, σηματοδοτεί μια νέα φάση για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και κυρίως για την ΚΑΠ. Ε, τέλος, η νομοθετική ευρωπαϊκή διαδικασία δίνει στο Κοινοβούλιο έναν αποφασιστικό ρόλο και ισότιμο ρόλο σε σχέση με το Συμβούλιο για την έγκριση των ε, προτάσεων της Επιτροπής. Χάρη στην απόφαση, το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να συνεισφέρει για να δώσει φωνή στην... Ε, να δώσει μεγαλύτερη φωνή στους πολίτες. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να ε, εγγυηθεί τις προσδοκίες μιας κοινωνίας προς μια βιώσιμη ανάπτυξη χάρη σε μια προσαρμοσμένη κοινή πολιτική στις ε, προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Σε ευχαριστώ για αυτή την, ε, τη δυνατότητα που μου δίνετε να κάνω αυτή την ε, εισαγωγή. Σηματοδοτώντας, σημειώνοντας κάποια στοιχεία που αναφέρει το κείμενο της Κομισιόν. Θα ξεκινήσει τώρα η συζήτηση στο σεμινάριο. Θα δώσω καταρχήν το λόγο τον Εσκίλ που είναι ο Σουηδός ε, Υπουργός ε, Γεωργίας. Εσκίλ. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά καταρχήν για την πρόσκληση σε αυτό το εργαστήριο μελέτης που λαμβάνει η χώρα τη σωστή στιγμή. Γιατί το θέμα αυτού του εργαστηρίου μελέτης αποτελεί θέμα μείζωνος σημασίας. Η κοινή γεωργική πολιτική και πώς αυτή θα διαμορφωθεί μετά το 2013 είναι ύψη προτεραιότητα και του Συμβουλίου. Διανύουμε μια ενδιαφέρουσα στιγμή λίγο πριν την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Κάτι που θα σημάνει τη στενότερη συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα αυτής της στενότερης συνεργασίας θα είναι πολύ επικοδομητικό και θα με βλέπετε όλο και πιο συχνά στο χώρο αυτό. Η συζήτηση για την ΚΑΠ μετά το 2013 βρίσκεται στις αρχές, βρίσκεται στα σπάργανά της. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έλαβε πρώτα η Γαλλική Προεδρία το φθινόπωρο του 2008 και κατόπιν η Ζεχική Προεδρία επικεντρώθηκε στις άμεσες ενισχύσεις. Εγώ θα αναφερθώ περισσότερο στο θέμα της ανάπτυξης της υπαίθρου. Θα γίνει μάλιστα μια ενημερωτική συζήτηση την επόμενη εβδομάδα για το θέμα αυτό. Κατά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών θα ζητήσω από τα κράτη-μέλη να εντοπίσουν τις ε, βασικές προκλήσεις που καλείται να αναλάβει η γεωργία και να αντιμετωπίσουν οι γεωργικές ζώνες. Πώς θα αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις. Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις σίγουρα είναι οι κλιματικές αλλαγές. Οι κλιματικές αλλαγές ε, είναι μια παγκόσμια πρόκληση και ίσως η σημαντικότερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει ο πλανήτης. Γιατί είναι πια εμφανείς αυτές οι κλιματικές αλλαγές. Στο άτυπο συμβούλιο του Βέξε στο Σεπτέμβριο, ήσουν εκεί άλλωστε Πάολο, μιλήσαμε για αυτό το θέμα της σχέσης κλίματος, υπεριβάλλοντος και γεωργίας και συμφωνήσαμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να διαδραματίσει κέριο ρόλο προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ταυτόχρονα για να προσαρμοστεί η γεωργία στις κλιματικές αλλαγές. Οι Ευρωπαίοι γεωργοί δίνανται και οφείλουν να συμμετέχουν περισσότερο στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και οι άλλοι τομείς της Ένωσης και καλό θα ήταν η Γεωργία να δώσει το καλό παράδειγμα. Επίσης θα πρέπει να συμπεριλάβουμε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικών αλλαγών στην κοινή γεωργική πολιτική όλο και περισσότερο. Όλα αυτά τα ζητήματα θα μας προβληματίσουν και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μην απομονώσουμε το θέμα του κλίματος. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η κοινωνία. Για παράδειγμα το θέμα της βιοπικιλότητας, το θέμα της διαχείρισης του ύδατος, που γίνεται όλο και πιο δύσκολη με τις κλιματικές αλλαγές. Οπότε οι κλιματικές αλλαγές και οι προκλήσεις τους θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού με τις υπόλοιπες προκλήσεις. Ένα άλλο θέμα που θα εξετάσουμε είναι το πώς ε, θα δώσουμε ενάψματα για τις οικονομικές δραστηριότητες στην Ήπεθρο. Το θέμα αυτό έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία μετά την ε, χρηματοπιστωτική κρίση της τελευταίας διετίας. Η Ήπεθρος, ε, οι αγροτικές ζώνες θα πρέπει να γίνουν ελκυστικές, δελεαστικές, να προσελκύουν τον κόσμο για να ασκεί εκεί τη δραστηριότητά του. Και οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα θα μας επιτρέψουν μία αύξηση των δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο. Επίσης θα προωθήσουμε μία δυναμική ανάπτυξη της Ήπεθρου. Να δώσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στην Ήπεθρο και σε αγροτικές ζώνες για να βοηθήσουν τις ζώνες αυτές να αναπτυχθούν. Η ΚΑΠ έχει ως πρωταρχικό της στόχο την αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων και προσπαθεί να δώσει μία απάντηση σε όλα αυτά τα προβλήματα. Σίγουρα υπάρχουν ελλείψεις στην ισχύουσα πολιτική και θα πρέπει από κοινού να βρούμε λύσεις για να τις ξεπεράσουμε. Κανείς δεν αμφισβητεί τη μεγάλη σημασία που έχει η κοινή αγροτική πολιτική και το ρόλο που διαδραμάτισε για την αποκατάσταση όρων θεμητού ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Χρειαζόμαστε μια γεωργική πολιτική που θα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα πολλές προκλήσεις και που θα είναι και δίκαιη για το φορολογούμενο. Σε ό,τι φορά τις άμεσες ενισχύσεις, υπάρχουν πολλές χώρες, ιδιαίτερα νέες χώρες μέλη, που ζητούν μία αλλαγή του συστήματος των άμεσων ενισχύσεων προκειμένου να εφαρμόζεται πιο δίκαια. Γιατί το σύστημα αυτό στηρίχθηκε σε μία ιστορική κατάσταση. Και αν κρατήσουμε τα ίδια αίτια αναφοράς και τα ίδια σημεία αναφοράς θα είναι αδύνατο να διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο. Θα πρέπει να γίνει μία μεγαλύτερη εξίσωση αυτών των άμεσων ενισχύσεων. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο της μελλοντική ΚΑΠ μετά το 2013. Επίσης, θα πρέπει να υλοποιήσουμε και τους στόχους αυτών των άμεσων ενισχύσεων. Να διαρωτηθούμε αν σήμερα οι άμεσες αυτές ενισχύσεις συμβάλλουν όντως στην υλοποίηση του στόχου των δίκαιων εισοδημάτων ή των αξιοπρεπών γεωργικών εισοδημάτων. Γνωρίζουμε ότι εξαιτία του συστήματος αυτού πολλές φορές αυξάνονται οι τιμέ των προϊόντων. Πολλές φορές ε, οι γεωργοί χρεώνονται για να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος παραγωγής. Όσοι τουλάχιστον θέλουν να αυξήσουν την παραγωγή τους. Και ως ε, Σουηδός Υπουργός Γεωργίας πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε εναλλακτικέ λύσει σχέση με το σύστημα άμεσων ενισχύσεων ή μάλλον να το τροποποιήσουμε για να θεραπεύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν ήδη σε ορισμένες περιοχές. Μία ενίσχυση που δίνεται άμεσα στον πολίτη και που δεν συμμετέχει η αγορά δεν ξέρω αν είναι λειτουργική. Για όλες τις προκλήσεις που σας ανέφερα προβλέπονται αυτές οι άμεσες ενισχύσεις στο δεύτερο πυλώνα. Αυτές είναι οι απόψεις μου για τη μελλοντική κοινή πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Εσκύλ. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σου. Φυσικά, μετά τις δύο πρώτες εισηγήσει θα γίνει μια συζήτηση. Γι' αυτό ετοιμάστε όλοι τις ερωτήσεις σας και τώρα θα δώσω το λόγο στη Μαριάν Φίσσαλμπολ. Ευχαριστώ, Μαριάν. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ καταρχάς που οργανώσατε αυτό το εργαστήρι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, ε, για το ότι μου δίνετε την ευκαιρία να πω δύο λόγια και εγώ με τη σειρά μου. Ε, ελπίζω που θα με συγχωρέσατε, που θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις πολύ εστιασμένα. Γιατί καταλαβαίνω ότι 10 λεφτά για να κάνω μια παρέμβαση για τη γεωργία δεν είναι αρκετά. Έχω πάρα πολλέ λεπτομέρειε να σα πω, γι' αυτό θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Θα ήθελα μόνος, καταρχά, μόνο καταρχά να ξεκαθαρίσω κάτι. Πιστεύω στεναρά ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρή ΚΑΠ για το μέλλον. Διάβασα διάφορα πράγματα για τις απόψεις μου, υποτίθεται, σε διάφορες εφημερίδες συχνά με περιγράφουν ως ε, υπερφιλελεύθερη που θέλει να τα αφήσει όλα στις αγορές, στο παιχνίδι των αγορών. Αυτό είναι βλακεία. Είναι ανοησίες, δεν αληθεύει. Και οποιοδήποτε έχει παρακολουθήσει τις συζητήσεις στις οποίες συμμετείχα, το ξέρει πολύ καλά. Ε, από την άλλη θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η κοινή αγροτική πολιτική Χρειάζεται περαιτέρω αλλαγέ για το μέλλον. Αλλά αυτές οι αλλαγέ θα πρέπει να τη δυναμώσουν και όχι να την αποδυναμώσουν. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει. Γιατί χρειαζόμαστε μια ισχυρή ε, πολιτική, αγροτική πολιτική και ισχυρή πολιτική ανάπτυξη πέθρου. Καταρχάς, λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν για την επισητιστική ασφάλεια. Ξέρουμε ότι ο πληθυσμός παγκόσμια αυξάνεται, αυξάνεται μέρα προς μέρα. Περιμένουμε από 7 δισεκατομμύρια σήμερα να φτάσει σε περίπου 9 δισεκατομμύρια ε, το 2050. Και ξέρουμε επίσης ότι τα μοντέλα, τα διατητικά, τα διατροφικά αλλάζουν. Παραδείγματος χάρη οι Ασιάτες τώρα αρχίζουν να τρώνε κρέας. Και όχι μόνο ρύζι. Και αυτό έχει επιπτώσεις βεβαίως. Επομένως, πρέπει να τονώσουμε την ε, γεωργική μας παραγωγή. Με βάση κάποιες εκτιμήσεις ε, πρέπει να αυξήσουμε τη γεωργική μας παραγωγή κατά 70 με 100% μέχρι το 2050. Η επισυντιστική ασφάλεια εξαρτάται μερικώς από το εμπόριο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να έχει μια θετική στάση προς, την, το εμπόριο γεωργικών αγαθών. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι βγάζουμε και λεφτά στο κάτω-κάτω από το εμπόριο. Από την άλλη, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την ε, εσωτερική μας παραγωγή και τη βάση που έχουμε για αυτή την παραγωγή. Εάν ένα μεγάλο τμήμα των ε, τροφίμων που παράγονται, παράγονται σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, υπάρχει μια φοβερή συγκέντρωση, τότε η προσφορά θα κινδυνεύσει. Θα είναι ευαίσθητη, θα εξαρτάται από κρίσεις, από κακό καιρό, από αρρώστιες. Δεν νομίζω ότι πρέπει να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν θα ήθελα να καταλήξουμε να είμαστε ευπαθείς σε ό,τι αφορά την παραγωγή τροφίμων. Όταν βλέπετε, ας πούμε, πόσο ευπαθείς είμαστε ε, κατά την εισαγωγή φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε κάποιους προμηθευτές που απλώς κλείνουν τους σωλήνες. Αν αυτό συνέβαινε στα τρόφιμα θα ήταν καταστροφικό. Δεν πρέπει λοιπόν να εκτεθούμε ε, σε άνθιο κίνδυνο. Δεύτερον, χρειαζόμαστε καλές πολιτικές για να έχουμε καλή διαχείριση της γης, και η γεωργία και η δασοκομεία καλύπτουν περίπου το 80% της ε, επικράτειάς μας. Και σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, αν αυτές οι γεωργικές ε, δραστηριότητες ξαφνικά σταματήσουν, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα ήταν ε, πάρα πολύ σοβαρές. Σε πολλές περιπτώσεις, η εγκατάλειψη της γης τάχιστα θα σήμαινε καταστροφή της γης και του εδάφους και ορισμένε περιοχές θα γίνουν απλούστατα έρημοι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περίπου το 1 τρίτο της γεωργικής μας γης είναι υψηλή αξίας. Είναι υψηλή βιοπικιλότητας, που απλώς χωρίς γεωργία θα καταστραφεί. Αυτή η βιοπικιλότητα θα χαθεί. Να μην ξεχνάμε ότι προσπαθούμε ε, ξεχνάμε υποτίθεται να σταματήσουμε την ε, επιδείνωση της βιοπικιλότητας μέχρι το, την επόμενη χρονιά. Επίσης, χρειαζόμαστε ισχυρή ΚΑΠ για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Περίπου το 9% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχονται από τη Γεωργία. Αυτό δεν είναι τεράστιο ποσοστό, αλλά παρόλα αυτά έχει μια σημασία. Όπως και άλλοι τομείς, ο γεωργικός τομέας θα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές του τα επόμενα χρόνια θα πρέπει επίσης να προσαρμοστεί στις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, τις οποίες αισθανόμαστε όλοι μας. Και τέλος, θα πρέπει να έχουμε μια ισχυρή ΚΑΠ για να υποστηρίξουμε ισορροπημένη ανάπτυξη των περιοχών της υπαίθρου. Σε ό,τι αφορά την πυκνότητα του πληθυσμού, οι αγροτικές περιοχές μας και η ύπεθρος είναι περίπου το 90% της επικρατείας μας συνολικά και φιλοξενεί περίπου το μισό του ευρωπαϊκού πληθυσμού, του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές από αυτές τις περιοχές έχουν τεράστιο δυναμικό. Είναι μέρη όπου μπορεί να ζήσει κανείς, να δουλέψει κανείς, αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βασικές υπηρεσίες, χρειάζεται δημόσια υποστήριξη για να ανθίσει αυτό το δυναμικό. Επομένως, αν χρειαζόμαστε ε, μια ισχυρή πολιτική τι μόρφη πρέπει να πάρει έτσι, μέσα σε, με γενικό τρόπο. Είμαι πραγματικά πεπισμένη ότι αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε πίσω. Να πάμε πίσω. Οι μέρες της βαριάς διαχείρισης τέλειωσαν, πέρασαν επιστρεπτοί. Κάθε πρόγραμμα έπαιξε το ρόλο του μια συγκεκριμένη ε, εποχή. Ούτω ή άλλω, ε, αυτή η προσπάθεια είχε αρνητικές αρνητικες παρενεργειε παρενέργειες και δεν υποστήριξε επαρκώ το εισόδημα των ε, γεωργών. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ή οποιοδήποτε πιστεύει ότι κάτι έχουμε, τέτοιο έχουμε στο μυαλό μας, νομίζω ότι κάνει λάθος. Ε, Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θέλω να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση, πλήρης απορρίθμιση. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι υπέρ των δημοσιονομικών περικοπών μόνο και μόνο για τις περικοπές για, ως αυτό σκοπό. Αντίθετα, θα πρέπει οι γεωργοί να μπορούν να ανταποκριθούν ανταγωνιστικά και εφάνταστα ε, με δημιουργικότητα στα σήματα της αγοράς θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις προσπάθειές του, ώστε η βάση παραγωγής μας να μην καταστραφεί. Μπορούμε να έχουμε ένα δίκτυο ασφαλείας, το οποίο δεν αποθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα. Και αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της γης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους γεωργούς μας με σεβασμό ως εταίρους που φροντίζουν το περιβάλλον. Οι ρυθμίσεις πρέπει να παίξουν το ρόλο τους, αλλά σε κάποιο βαθμό θα πρέπει να βοηθήσουμε τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν το κόστος της ε, φροντίδας του περιβάλλοντος. Γιατί το κόστος αυτό σπάνια το πληρώνει η αγορά ή δεν το πληρώνει καθόλου. Θα μπορούσα να πω το ίδιο και για την ε, κλιματική αλλαγή. Και εδώ οι ρυθμίσεις και οι κανόνες έχουν το ρόλο τους. Αλλά αν ε, καταστρέψουμε τους γεωργούς μας με κανόνες χωρίς να σηκώσουμε το χεράκι μας για να τους βοηθήσουμε. Απλώς θα μεταφέρουμε την ε, παραγωγική μας ε, βάση και το παραγωγικό μας δυναμικό στο εξωτερικό. Και πάλι τελικά θα εξαρτώμεθα από τις εισαγωγές. Θα πρέπει επίσης να εξηγήσουμε μετά στο κοινό γιατί δημιουργούμε περισσότερες, ε, περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου εισάγοντας τρόφιμα τα οποία παράγονται με περιβαλλοντικά πρότυπα σαφώς κατώτερα από αυτά που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι επενδύσεις, ούτω ώστε το σύστημα το αγροτικό να είναι πιο φιλικό προς το κλίμα μέσω της τεχνολογίας, κατάρτισης και μερικές φορές μέσω απλών αλλαγών. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ ε, σόφρονη επένδυση. Σε ό,τι αφορά τις ε, γενικότερες ε, παγκόσμιες εξελίξεις, νομίζω ότι η βασική μας προσέγγιση του να έχουμε μια παλέτα από μέτρα μέσα από τα οποία τα κράτη-μέλη ε, και οι περιοχές μπορούν να διαλέξουν ό,τι τους βολεύει και το ό,τι τους συμφέρει και τους ταιριάζει, νομίζω είναι μια πολύ σωστή προσέγγιση. Είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να ανασκουμποθούμε και να βελτιώσουμε την ΚΑΠ. Φυσικά για την ΚΑΠ ε, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να πετάξουμε αυτά τα πράγματα τα οποία δούλεψαν στο παρελθόν αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να γίνουμε και όμοιροι της ιστορίας και του παρελθόντος. Ένα τελικό σχόλιο. Το να κερδίσουμε και να κρατήσουμε την υποστήριξη για την ΚΑΠ σημαίνει ότι έχει σαφείς στόχους, τους οποίους μπορεί να δεχτεί το κοινό, να τους καταλάβει και να τους δεχτεί. Ε, σαφείς, λογικούς στόχους, που βεβαίως μπορεί να έχουν επιπτώσεις για το πώς μοιράζονται τα κράτη μεταξύ των κρατών μελών. Ο Σουηδός υπουργό ε, μίλησε για αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα το πώς θα μοιράσουμε τα λεφτά μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, το ξέρω. Και φυσικά θα πρέπει να είμαστε πολιτικά ρεαλιστές εδώ. Αλλά θα πρέπει να είμαστε επίσης και πολιτικά ρεαλιστές με, με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή δεν μπορούμε από τη μία να υπερασπιζόμαστε την ΚΑΠ βασική και ζωτική κοινοτική πολιτική, αν από την άλλη ο κόσμος θεωρεί ότι η συζήτηση ε, εστιάζεται στο πώς θα κρατήσει ο καθένας το δικό του μερίδιο, θα αυξήσει το μερίδιο της πίτας. Νομίζω ότι μπορούμε να κερδίσουμε το επιχείρημα ε, για την κοινή αγροτική πολιτική. Μπορούμε να πείσουμε το κοινό ότι μπορεί να παίξει ένα ζωτικό ρόλο για την πράσινη ανάπτυξη που χρειαζόμαστε για το μέλλον. Επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, να κάνω ένα σύντομο σχόλιο για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού και για το κείμενο αυτό που μιλούσε για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού, που δεν υπάρχει. Στην πραγματικότητα, όταν, το άκουσα, όταν άκουσα για αυτό το έγγραφο, εξεπλάγινε. Εγώ δεν το είδα ποτέ αυτό το κείμενο. Νομίζω ότι είναι κάποιοι πάλι τη Κομισιόν, οι οποίοι γράφανε, ας πούμε, τις δικές τους ιδέες για το τι θα μπορούσε να είναι το μέλλον. Από δημοσιονομικής πάντα πλευράς. Αυτό το έγγραφο είναι ήδη στον κάλαθο των αχρήστων. Και η επόμενη επιτροπή θα παρουσιάσει το δικό της έγγραφο. για τη μελλοντική αναθεώρηση του προπολογισμού. Όταν το είδατε, ε, όταν είδατε τι έγραφε για την ε, συγχρηματοδότηση, ελπίζω να καταλάβατε ότι αποκλείεται να είναι δικά μου αυτά τα, αυτές οι ιδέες. Γιατί ξέρετε πολύ καλά τι πιστεύω για την συγχρηματοδότηση. Σας λέω επίσημα, πιστέψτε με, αυτό το έγγραφο δεν υπάρχει και σε καμία περίπτωση δεν θα τεθεί επιτάπητος, αλλά όμως η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις απόψεις της για το θέμα του προπολογισμού. Δεν μπορώ τώρα να, σας, να προδικάσω με τι θα μοιάζει αυτή η συζήτηση για τον προπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αγαπητή Μαριάννα, με αυτό το χειροκρότημα απελευθερώνεται ο κόσμος. Ε, αυτό σημαίνει ότι μας άρεσε η παρέμβασή σου. Σε ευχαριστούμε γιατί διευκρίνησες ε, ότι αυτό το έγγραφο δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά εγώ το είδα στις πρώτες σελίδες των πιο σημαντικών εφημερίδων. Γι' αυτό ανησύχησα πάρα πολύ, όχι μόνο εγώ, όλοι μας. Σε ευχαριστούμε λοιπόν για την παρέμβασή σου και σε ευχαριστούμε για αυτή τη διευκρίνηση. Η οποία μας ενθουσίασε και μας ανακούφισε. Και τώρα μπαίνουμε στο ψητό του σεμιναρίου. Όπως ξέρετε έχουμε τέσσερις εμπειρογνώμονες ε, που, γνωρίζουν, που είναι πολύ γνωστοί, ε, ο καθένας στον τομέα του. Ε, θα δώσουμε το λόγο στους δύο πρώτους εμπειρογνώμονες, τον καθηγητή Μπάκουελ από το Country Land and Business Association και συνεχεία στον κύριο Σατελιέ από την Ίνερα. Και συνεχεία θα ξεκινήσει η συζήτηση. Γι' αυτό Έχουμε μία πρώτη συζήτηση με τις δύο πρώτες παρεμβάσεις, μετά συζήτηση και μετά τις επόμενες δύο παρεμβάσεις. Τώρα, με μεγάλη χαρά, θα δώσω το λόγο στον ε, καθηγητή κύριο Μπάκουελ. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία αυτή να απευθυνθώ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα αυτή τη μοναδική στιγμή όπου το Κοινοβούλιο πρόκειται να λάβει πλήρη στην απόφαση. Και γι' αυτό λοιπόν η σημασία του είναι ακόμη πιο μεγάλη από ότι στο παρελθόν. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι η ΚΑΠ βρίσκεται σε φάση μεταρρυθμιστική ουσιαστικά από τότε που ξεκίνησε. Είτε θεωρούμε ότι ξεκίνησε το 65 είτε το 68 δεν έχει σημασία και η ΚΑΠ ε, κατά ευφύ τρόπο πάντα προσαρμοζόταν στην πολιτική και οικονομική και κοινωνική κατάσταση που, προ... που άλλαζε και αυτή στην ε, Ευρώπη. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι από το 1992 όταν η παλιά ΚΑΠ η οποία ήταν αποκλειστικά υποστήριξη των τιμών στην αγορά από τότε λοιπόν, από τότε που το σύστημα αυτό μεταρρυθμίστηκε ή ξεκίνησε μάλλον η μεταρρυθμιστική διαδικασία, μα ξέρει, υπήρξε μια τάση μεταρρύθμισης διαρκής. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αλλάζει η ΚΑΠ. Αυτό που δεν είναι σαφές είναι τι μορφή παίρνει και γι' αυτό λοιπόν η συζήτηση που διεξάγεται τώρα και που θα διεξαχθεί στο μέλλον θα καθορίσει ε, τη μελλοντική αυτή μορφή της ΚΑΠ μετά το 2013. Και θα πρέπει να εστιαστούμε λοιπόν στη συζήτηση αυτή στο μεγαλύτερο τμήμα της ΚΑΠ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις δημόσιες δαπάνες, που είναι το ενιαίο πληρωμών. Και σε αυτό θα εστιάσω και τις παρατηρήσεις μου. Το πρόβλημα είναι ότι οι αποδέκτες των πληρωμών αυτών θεωρούν ότι είναι ε, μόνιμο το εισόδημα αυτό, ενώ όλοι οι υπόλοιποι είναι σε φάση σύγχυσης και θεωρούν ότι είναι μάλλον ένα προσωρινό σύστημα βοήθειας. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια συμφωνία μεταξύ των αποδεκτών και της υπόλοιπης κοινωνίας, γιατί αυτή η αβεβαιότητα για τις πληρωμές δεν είναι καλή για κανέναν, ούτε για την Ευρώπη και τις πολιτικές της, γιατί δέχεται κριτικές από όλους ε, εκτός του αγροτικού τομέα και από όλους εκτός ε, της Ευρώπης. Ούτε για τους γεωργούς είναι καλή η κατάσταση αυτή γιατί βρίσκεται υπό διαρκή αμφισβήτηση το εισόδημά τους. Δεν υπάρχει βεβαιότητα. Θα πρέπει να μην προστίθεται επιπλέον αβεβαιότητα. Και γι' αυτό λοιπόν γίνεται η όλη συζήτηση. Ήταν πολύ ενδιαφέρον που ακούσαμε τον πρόεδρο της Επιτροπής και την Επίτροπο πώς περιγράφουν αυτό το έγγραφο της ε, Επιτροπής, το οποίο είναι ανεπίσημο, αλλά ωστόσο υπάρχει και υπάρχουν επιχειρήματα ότι θα πρέπει να περιοριστεί θα περιοριστούν οι δαπάνες για την ΚΑΠ και συμφωνώ απόλυτα από αυτά που ακου... με αυτά που ακούστηκαν ότι η περικοπή των δαπανών, των κονδυλίων και μετά η συζήτηση για την ανακατανομή και η μετέπειτα συζήτηση για την μεταρρύθμιση του είναι ο κόσμο, αν θέλετε ανάποδα. Είναι αντίστροφο από αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Πρώτα θα πρέπει να συζητήσουμε του στόχου της ε, πολιτική, να δούμε τι θέλει ο κόσμο, τι, θέλουν, τι θέλει ο κλάδος και πώ πρέπει να μεταρρυθμίσουμε τον κλάδο και όταν θα έχουμε συμφωνήσει επί των στόχων, τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε την ανακατανομή των πόρων και να δούμε κατά πόσο επαρκούν και συμβάλλουν στην συνοχή και μόνο τότε έχει νόημα να αποφασίσουμε για το κλάσμα των δημοσίων δαπανών που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για να υποστηρίξουμε την πολιτική αυτή. Και υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος σε περίπτωση που ξεκινήσουμε αντίστροφα από το τέλος. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος ε, της πολιτικής αυτής μετά το 2013 και φυσικά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις, ε, τις ε, υποχρεώσεις που ορίζονται στη συνθήκη. Αλλά αυτό που προτείνει να σκεφτείτε είναι το εξής. Το σλόγγαν που χρησιμοποιείται είναι το σλόγγαν των τροφίμων και της περιβαλλοντικής ασφάλειας. Και αυτά τα λόγια τα άκουσα και στα λόγια της Επιτροπής και στα λόγια του Προέδρου της Επιτροπής Γεωργικών Υποθέσεων. Υπάρχει ανάγκη να δοθούν τρόφιμα στον κόσμο βάσει καλλιεργήσιμων γεών, οι οποίες απειλούνται από την αλλαγή του κλίματος, απειλούνται και οι υδατινοί πόροι. Αλλά υπάρχει και η πρόκληση της ε, κάλυψης των διτροφικών μας αναγκών, το οποίο φυσικά θα πρέπει να καλυφθεί ως ανάγκη, αλλά παράλληλα και της προστασίας του εδάφους, των υδάτων και της τοποθεστών ε, του περιβάλλοντος. Και όλα αυτά φυσικά αυτές οι δύο προκλήσεις είναι αλληλένδετες, γιατί η παροχή τροφίμων εξαρτάται από το περιβάλλον και το περιβάλλον εξαρτάται από τις δομές και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε. Και το θέμα είναι το εξής αν τα συμφέροντα, τα περιβαλλοντικά και τα γεωργικά δεν ε, συνδυαστούν για να ενταχθούν στα πλαίσια της δεύτερης γραμμής του προϋπολογισμού, νομίζω, αν δεν συνδυαστούν μάλλον, εκεί δεν θα συνδυαστούν πουθενά. Και νομίζω ότι είναι πολύ γερή η βάση που αποδεικνύει το γεγονός αυτό. Για να επικεντρωθούμε τώρα πιο συγκεκριμένα. Αν θέλουμε να γίνει μια λεπτομερή συζήτηση για την ε, τροποποίηση της ΚΑΠ για να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις θα ήταν βασικά να κοιτάξουμε, χρήσιμο να κοιτάξουμε ποια είναι, ποιες είναι οι αδυναμίες του τρέχοντος συστήματος. Κάποιοι ίσως πούν ότι δεν υπάρχουν αδυναμίες. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Υπάρχουν δύο βασικά προβλήματα με τη σημερινή ΚΑΠ, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όσο έχουν. Καταρχάς, η νομιμότητα των ενιαίων πληρωμών και τα θέματα που αφορούν την ε, παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών, όπως τα αποκαλώ εγώ. Τι εννοώ με την νομιμότητα της ενιαίας πληρωμής, γιατί είναι κάτι το σοβαρό φυσικά αυτό. Μιλάμε για το 75% των συνολικών δαπανών σήμερα. Το πρόβλημα είναι ότι οι ακαδημαϊκές μελέτες κοιτώντας τις λεπτομέρειες των πληρωμών αυτών για το ποιος τις προσλαμβάνει και γιατί τις χρησιμοποιεί, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος. Ενισχύουν ε, το εισόδημα, κάποιοι μιλούν για σταθεροποίηση, κάποιοι άλλοι αναφέρουν ότι ε, σχετίζεται με τα πρότυπα, τα περιβαλλοντικά και τα της εφημερίας των ζώων. Κάποιοι άλλοι λένε ότι οι αγρότες παρέχουν υπηρεσίες περιβαλλοντικές. Άλλοι μιλούν για επιστημιστική ασφάλεια. Όλα αυτά τα επιχειρήματα έχουν κάποια ουσία, αλλά δεν επαρκούν για να εξηγήσουν το ποσό που δίνουμε στους αγρότες. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Επί της αρχής λοιπόν υπάρχει μια ουσιώδης ε, δυσκολία σε ό,τι αφορά το σύστημα άμεσων πληρωμών. Και στην πράξη επίσης υπάρχει πρόβλημα, γιατί στην πράξη αρκούν τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε για να δούμε πόσο μεγάλη είναι η εξάρτηση των εκμεταλλεύσεων από τις πληρωμές αυτές. Από τις ε, πληρωμές αυτές. Το ποσοστό των άμεσων πληρωμών είναι από 1% έως 106% και κατά μέσο όρο 35%. 35% δηλαδή των εκμεταλλεύσεων εξαρτάται από αυτές τις πληρωμές. Άρα όσοι υποστηρίζουν την κατάργησή τους και πολλοί την υποστηρίζουν θα πρέπει να εξηγήσουν πώς θα γίνει η μεταρρύθμιση του συστήματος για να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι και η κατανομή στο ιστορικό των κρατών μελών είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολη. Κοιτώντα ε, την εξάρτηση βλέπουμε ότι σε κάποιες περιοχές είναι στα βοσκοτόπια για παράδειγμα, είναι πάνω από 100% αυτή η εξάρτηση και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τους αγρότες, για τους ε, εκτροφείς, γιατί εξαρτώνται από, μια, ε, από ένα σύστημα το οποίο βρίσκεται διαρκώς υπό αμφισβήτηση. Και ξέρουμε ότι αυτό γίνεται ενδεχομένως ανά εκτάριο, ανά αποδέκτη. Και πάλι, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ποιοι είναι οι στόχοι της ΚΑΠ αυτά τα προβλήματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Το δεύτερο βασικό πρόβλημα έχει να κάνει με τα περιβαλλοντικά αγαθά, με τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, γιατί η διαχείριση των γεών πολύ απλά δεν τα πηγαίνει καλά. Το πρόβλημα είναι το εξής. Η κοινωνία δίνει τεράστια αξία σε αυτές τις υπηρεσίες οικοσυστήματος, τις οποίες μπορούν να παρέχουν μόνο οι αγρότες και οι εκτροφείς. Και πολύ απλά δεν αποδίδουν επαρκώς. Να προειδοποιήσω ότι ο όρος δημόσιο αγαθό θα μας οδηγήσει σε προβλήματα εάν δεν υπάρχουν ποσοτικοποιήσεις και συγκεκριμένοι ορισμοί. Η διάγνωση λοιπόν των προβλημάτων αυτών προδιαγράφει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι μεταρρυθμίσεις. Πιο πολύ δηλαδή η κατεύθυνση που ακολουθούμε από το 1992 να αντιμετωπίσουμε τα συστήματα, τα στοιχεία αποτυχίας της αγοράς παρά να προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις αγορές. Και αυτό που λείπει είναι η βοήθεια η οποία είναι απαραίτητα, απαραίτητη για να υποβοηθήσουμε την μεταρρύθμιση της, ε, του γεωργικού κλάδου και αυτό είναι κάτι το απαραίτητο. Όλοι οι κλάδοι πρέπει να μεταρρυθμίσονται, δεν μπορεί να ξέρουμε την γεωργία. Άρα, ας κάνουμε την ανάγκη φιλότιμο. Εφόσον θα υπάρξουν περικοπές στις πληρωμές αυτές, αυτό το καθορίζει ε, ο προπολογισμό και άλλωστε και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν, δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι που θέλουμε, ας φροντίσουμε τουλάχιστον να κινηθούμε προς την κατεύθυνση που επιθυμούμε. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω στην ΚΑΠ του 2013 να περιλαμβάνονται τα πέντε εξή στοιχεία. Το βασικό είναι ότι οι ενιαίες πληρωμές, ακόμα και να αλλάξουμε τον τίτλο και την ονομασία, ας, ας πούμε για παράδειγμα μεταβατικές ρυθμίσεις, τι θα κάνουν. Θα παραμείνουν ένα σύστημα του παρελθόντος, όχι του μέλλοντος. Ας το πούμε ότι πρόκειται για μία προσωρινή βοήθεια προσαρμογής, γιατί η προσαρμογή στην αλλαγή είναι κάτι το πολύ έξυπνο στην Ευρώπη. Αν μπορέσουμε λοιπόν με τα χρήματα αυτά να βοηθήσουμε τους αγρότες να μεταρρυθμιστούν, να αλλάξουν το σύστημά τους, νομίζω ότι θα έχουμε σημαντικά ωφέλη. Δεν θα αναφέρω τα υπόλοιπα συστήματα, τα υπόλοιπα στοιχεία, γιατί θα αναφερθούν και σε μελλοντική παρουσίαση, σε μια επόμενη παρουσίαση. Στο D βλέπουμε ότι οι αποκεντρωμένες περιοχές της Ευρώπη αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα γιατί εκεί είναι η μεγαλύτερη εξάρτηση από τις πληρωμές και θα πρέπει να δίνονται, να παρέχονται οι πληρωμές αυτές με σωστό τρόπο για να πετύχουμε τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Για παράδειγμα, την ε, πρόληψη των πλημμύρων και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να τεθεί ο στόχος για τις περιοχές αυτές. Αν προσπαθήσουμε να συνδέσουμε τις ιδέες αυτές με τις τρέχουσες πολιτικές, θα διαπιστώσουμε ότι οι μελλοντικέ λύσεις εντάσσονται ουσιαστικά στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα. Έχουν τέτοια χαρακτηριστικά, δηλαδή μία προσέγγιση προγραμματισμού όπου τα κράτη-μέλη επιλέγουν στο βαθμό, το βαθμό που θέλουν να ακολουθήσουν τα μέτρα που προτείνονται. Το βασικό πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση και εδώ μου τελειώνει και ο χρόνος. Θεωρώ ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε να δώσουμε πιο πολλά τέτοια αγαθά στον πρωτοπυλώνα, είτε χρησιμοποιώντας με πιο ευρύ τρόπο το άρθρο 68, αλλά θεωρώ ότι αυτό δεν είναι σωστό, δεν είναι έξυπνο, γιατί πιο πολύ ταιριάζει ο, ο δεύτερο πυλώνα. Το βασικό, το κρίσιμο πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση. Και ξέρουμε ότι τα βασικά προβλήματα που σχετίζονται με χρηματοδότηση είναι κατά πόσο μιλάμε για πιο πολύ modulation ή κατά πόσο μιλάμε για την ανακατανομή των ορφών σε ό,τι αφορά την ενιαία, της ενιαίας πληρωμής. Η απάντηση μάλλον αποτελεί κάτι το ενδιάμεσο, αλλά το βασικό είναι το εξή. Όταν θα κινηθούμε προς το δεύτερο πυλώνα, για να έχουμε δηλαδή προγράμματα τύπου δεύτερου πυλώνα, θα πρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι σε ό,τι αφορά τη συγχρηματοδότηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι συνολικέ δαπάνε για την ΚΑΠ δεν μπορούν να αυξηθούν. Και εδώ ακούγονται πάρα πολλέ φωνέ για τον περιορισμό των δαπανών αυτών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορούν να αυξηθούν. Άρα, για να μεταφερθούν τα κονδύλια από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα και να ζητήσουμε και επιπλέον κονδύλια, πολύ απλά δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθεί με καλύτερο τρόπο η συγχρηματοδότηση. Να το θέσω αλλιώ. Αν θέλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τους ε, σκοπούς της ΚΑΠ, ας ε, μοιράσουμε τα κονδύλια μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα, για να μην δεσμευτούμε από τις υφιστάμενες δομές. Ιδάλλως, πολύ φοβάμαι ότι θα περάσουμε τα επόμενα δύο χρόνια ε, με το να διαφωνούμε για το πώς θα πρέπει να ανακατανύμουμε τα, τις δαπάνες στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα. Να κλείσω λέγοντας ότι δεν πρέπει να μπούμε σε υπερβολικές λεπτομέρειες για το πρώτο και το δεύτερο πυλώνα. Γιατί αυτό απασχολεί μόνο τον κλάδο το γεωργικό και ακόμα δυσκολευόμαστε να πείσουμε τον κόσμο γιατί χρειάζεται αυτό το 0,5% του κοινοτικού ΑΕΠ για να χρηματοδοτήσουμε αυτό τον κλάδο. Πρόκειται για μια ιστορική ευκαιρία για το Ευρωκοινοβούλιο να συνδράμει σε αυτή τη ε, διαδικασία μεταρρύθμισης προκειμένου να αλλάξει αυτή η ροή, να αλλάξει αυτή η κριτική σε κάτι το οποίο μας κάνει περήφανος. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας και τώρα πριν να ξεκινήσει μια σειρά παρεμβάσεων που έχουμε ήδη προβλέψει, θα δώσω το λόγο στον κύριο, στον κύριο Σάτελιε από το Εθνικό Ινστιτούτο Αγρονομικής Έρευνας, το ΙΝΡΑ. Merci, Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που λαμβάνω το λόγο σε μια τόσο ταραγμένη εποχή της Ευρωπαϊκής Γεωργίας που έρχεται αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις. Θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί προς τις μελλοντικέ λύσεις, να μην είμαστε αδιάλακτοι και κλειστοί και να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε πολλά πράγματα. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Εγώ θα ασχοληθώ περισσότερο με τους μηχανισμούς ρύθμισης των αγορών. Πιστεύω ότι η ΚΑΠ αντιμετωπίζει τρεις ε, βασικές και πρόσφατες ε, εξελίξεις. Μια μεγάλη ρευστότητα των τιμών, άνευ προηγουμένου, και αυτή η αστάθεια των τιμών δεν ε, επηρεάζει μόνο την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά τη σχέση της ΚΑΠ με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, μέσω κυρίως των διαπραγματεύσεων στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Γνωρίζουμε ότι μία από τις ε, ιδέες που είχαν πριτανεύσει στη Συμφωνία του Μαρακέ είναι ότι η φιλελευθερωποίηση έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά και κάποιες ανεπάρκειες. Και φυσικά η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε την τελευταία δεκαετία να καταλήξουμε σε συμφωνία στο γύρο της Δόχα δείχνει πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθούμε ως προς τα ευεργετήματα τη απόλυτη απελευθέρωση των γεωργικών αγορών, ιδιαίτερα στι σχέσει μα με τι αναπτυσσόμενες χώρε. Δεύτερο σημαντικό θέμα που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι υπάρχει πίεση για τον προπολογισμό τη ΚΑΠ, δυστυχώ, ε, Γιατί πολλοί γεωργοί, όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και στην Ισπανία και τη Γαλλία, πολλοί γεωργοί δεν θα έχουν την πολυτέλεια να αντιμετωπίσουν μία ΚΑΠ που θα είναι υπερβολικά απαιτητική και θα συρρυκνώνεται ο προπολογισμό της. Πιστεύω ότι έτσι θα έρθουν σε πολύ δύσκολη θέση πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, και ίσως και να συνθλιβούν. Αυτή είναι η δύσκολη κατάσταση που διανύουμε σήμερα και θα πρέπει να είμαστε πολύ συνετοί ε, και να μην πετάμε στα, στα, στα καλάθια των αχρήστων πριν εξετάσουμε καν ορισμένες εκθέσεις. Το ίδιο ισχύει ε, και με τους γεωργικούς που αν φοβούνται το μέλλον δεν πρόκειται ούτε να επενδύσουν ούτε να εγκατασταθούν στις αγροτικές ζώνες. Και ίσως έτσι πληγεί η κοινή γεωργική πολιτική επειδή θα είναι αδιαφανής και μεσοπρόθεσμα. Γι' αυτό και είναι απαραίτητη η σημερινή συζήτηση. Πολλοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι ο γεωργικός τομέας είναι ένας ιδιάζων τομέας που χρήζει και στο μέλλον θα χρειάζεται ακόμη την κρατική παρέμβαση, γιατί εκφίσως οι γεωργικές αγορές είναι ασταθείς, ε, ε, επηρεάζεται η προσφορά από τις κλιματικές καταστάσεις, είναι βραχυπρόθεσμα ανελαστική και είναι κάτι που ισχύει, ισχύει στο παρελθόν, θα ισχύσει και στο μέλλον. Γι' αυτό και θα το διαπιστώσουμε πολλές φορές και στο μέλλον. Βέβαια, οι γεωργοί ε, γνωρίζουν την κατάσταση του κίνδυνου, αλλά δεν τους αρέσει ο κίνδυνος. Και όσο αισθάνονται τον κίνδυνο, επενδύουν όλο και λιγότερο. Αν αισθάνονται μια ασφάλεια, θα επενδύσουν περισσότερο. Και αναφέρεται και η, ε, η παραγωγή των αγοραίων αγαθών ε, σε σχέση με τις ε, κρατικές δημόσιες πολιτικές. Κάτι που δεν αναφέρουμε στην Ευρώπη είναι ότι η γεωργία ε, συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης σε διεθνές επίπεδο. Και η σχέση μεταξύ της ΚΑΠ και των υπόλοιπων χωρών είναι κάτι που θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και να μην το ξεχνούμε στη συζήτηση που γίνεται σε κοινοτικό επίπεδο. Ένα άλλο σημείο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι η γεωργία είναι ένας τομέας που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται στρατηγικός, παρόλο που το θέμα των εμπάργων δεν είναι τόσο στη μόδα σήμερα όπως το παρελθόν άλλο που είδαμε είναι ότι η ΠΑΚ εξελίχθηκε πάρα πολύ από το 1992. Και για να θέσουμε σε τροχιά τη μελλοντική ΚΑΠ, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη μας σε μια δεκαπενταετία σταδιακής προσαρμογής της ΚΑΠ, που είχε κάποιες ανεπάρκειες, όπως είπα, αλλά είχε και πολλά πλεονεκτήματα. Και στην συζήτηση που θα έχουμε, δεν θα πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη μας στη μεταρρυθμιστική διαδικασία. Ένα άλλο σημαντικό θέμα, γιατί το έγγραφό μου αφορά κυρίως ε, τη ρύθμιση των αγορών, είναι ότι μετά από μία δεκαπενταετία σταδιακών μεταρρυθμίσεων της ΚΑΠ, διαπιστώνουμε ότι η ρύθμιση των αγορών ε, έχει, ε, ε, αντιπροσωπεύει ένα μικρό τμήμα του προπολογισμού τη ΚΑΠ σήμερα, σε αντίθεση με τι αποσυνδεδεμένε ενισχύσει. Γιατί η ρύθμιση των αγορών είναι το 8% των δαπανών τη ΚΑΠ. Επίσης, οι εξαγωγικές επιστροφές ουδέποτε δεν ήταν τόσο χαμηλές όσο σήμερα. Και η αποθεματοποίηση έχει πιο περιθωριακό χαρακτήρα. Οπότε ουσιαστικά γυρίσαμε την πλάτη σε μια γεωρική πολιτική που πολλές φορές ήταν αφιλεγόμενη σε ό,τι αφορούσε τις εξαγωγικές επιστροφές, αλλά σήμερα δεν αφισβητείται κάτι τέτοιο και έχει περιοριστεί ως προς αυτό. Γιατί? τα μέτρα και τους μηχανισμούς ρύθμισης. Καταρχήν, να πούμε δύο λόγια για τους τελωνιακούς δασμούς. Λέμε γενικώ ότι οι τελωνιακοί δασμοί είναι ένα κέρδος για τους παραγωγούς, μία ζημιά για τους καταναλωτές, αλλά είναι σε τελική ανάλυση ένα κέρδος για τους φορολογούμενους. Κάθε φορά που μειώνουμε τις ελληνικούς σταθμούς από το Μαρακές, έχουμε επιτρέψει κάποιες άμεσες ενισχύσεις. Οπότε για το φορολογούμενο θα πρέπει να θέσουμε τη συζήτηση με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και όρους. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό στις συζητήσεις είναι ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και η ανάλυση της επίπτωσης της μείωσης των τελωνιακών δασμών για την Γεωργία είναι κάτι πολύ περίπλοκο. Γιατί υπάρχουν πολλά σημεία που είναι αλληλένδετα. Πολλά εξαρτώνται από την ε, ιδιάζουσα κατάσταση κάθε προϊόντος. Να μην έχουμε ενοποιημένους ε, δασμούς ε, και εφαρμοσμένους δασμούς. Να μην υποτιμούμε το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές ορισμένων γεωργικών προϊόντων αυξάνονται και θα συνεχίσουν να αυξάνονται στο μέλλον. Αυτά προβλέπουν ορισμένοι οργανισμοί πρόγνωση, ενώ οι ευρωπαϊκέ τιμέ έχουν μειωθεί. Α μην ξεχνούμε και του μη δασμολογικού φραγμού. Άλλωστε στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να, αναλύουμε, να ξεχνούμε όταν αναλύουμε τη δασμολογική προστασία την αυτοπροστασία που εφαρμόζουν οι ίδιοι οι καταναλωτές που προτιμούν να καταναλώνουν ντόπια προϊόντα και όχι εισαγόμενα. Η Επιτροπή Γεωργίας της ΠΟΕ από το Δεκέμβριο του 2008 προβλέπει μία μείωση, μέση μείωση του, του τελωνιακού δεσμού κατά 54%. 4% για τα ευαίσθητα προϊόντα. Έχουμε μια ιδιάζουσα λοιπόν κατάσταση, κυρίω για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Τώρα, ποια στρατηγική θα εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στι προτάσει τη Επιτροπή Γεωργία του ΠΟΕ. Η πρώτη ιδέα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι όλα τα προϊόντα ευαίσθητα ως προς την μείωση των τελωνιακών δασμών. Επίσης θα πρέπει να δεχθούμε την ιδέα ότι ορισμένες χώρες και κυρίως ε, οι αναπτυσσόμενες χώρες θα μπορέσουν να προστατεύσουν την παραγωγή τους, όχι μειώνοντας τα, τους τελωνιακούς δασμούς, αλλά ίσως αυξάνοντας τους για να προστατεύσουν την, τοπική τους, ε, την τόπια τους παραγωγή. Ακόμη και δεν είναι ανταγωνιστικέ απέναντι στη μαζική ευρωπαϊκή παραγωγή. Επίση, ε, τα λίγα ευαίσθητα προϊόντα που έχουμε θα πρέπει να τα κατευθύνουμε στην ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή, που καταλήγει σε μία γορέα προϊόντα. Για παράδειγμα, βόλιο κρέας και ίσως γαλακτοκομική παραγωγή. Κυρίως όμως ε, παραγωγή βόλιο κρέατος που δεν μπορεί να αντέξει τον ανταγωνισμό της Βραζιλίας για παράδειγμα ή άλλων χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ελλείμματα σε ορισμένες παραγωγές, στο πρόβιο κρέας για παράδειγμα. Αλλά αν γίνει ελληματική και για το βόλιο κρέας θα διευκολυνθεί η αποδοχή όλο και μεγαλύτερων εισαγωγών από άλλες χώρες. Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγικές επιστροφές, ουδέποτε δεν ήμασταν τόσο κοντά στην κατάργησή τους. Γιατί όλοι ξέρουν από το 2008 δεν ξοδέψαμε ούτε ένα δισεκατομμύριο ευρώ για τις εξαγωγικές επιστροφές. Και μάλιστα μας ευνόησαν στο σημείο αυτό πολύ υψηλέ διεθνείς τιμές για ορισμένα προϊόντα. Πάντως, ο μηχανισμός αυτός των εξαγωγικών επιστροφών θα χαθεί αργά ή γρήγορα που είναι χρήσιμο σε περίπτωση της κρίσης, αλλά εδώ και 15 χρόνια η, πολιτική, η γεωργική πολιτική προσαρμόζεται προκειμένου να απαλλαχθεί κάποια στιγμή από τις εξαγωγικές επιστροφές και νομίζω τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την κατάργησή τους. Αυτές οι εξαγωγικές επιστροφές θα πρέπει να καταργηθούν. Ούτως ή άλλως αφισβητούνται από πολλές χώρες και μη κυβερνητικές οργανώσεις και στον ΠΟΕ. Και σε τελική ανάλυση το διακύβευμα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να εξαγάγουν χωρίς εξαγωγικές επιστροφές τα προϊόντα τους. Και μην ξεχνάτε και τη συναλλαγματική ισοτιμία, που βρίσκεται και στο επίκεντρο της συζήτησης. Δεν θα πρέπει να αποσυνδέουμε την νομισματική πολιτική από τη γεωργική πολιτική. Και το γεγονός ότι υπάρχει ένα ισχυρό ευρώ απέναντι στο δολάριο αποβαίνει εις βάρος ε, των εξαγωγών μας και μας οδηγεί στην χρήση των εξαγωγικών επιστροφών. Σε ό,τι αφορά τις εγγυημένες τιμές, στα δίκτυα ασφαλείας, νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα των ελάχιστων αποθεμάτων για τα προϊόντα που επιδέχονται αποθεματοποίηση, για παράδειγμα τα σιτηρά. Και ίσως θα πρέπει στα διεθνή βήματα να ευαθύνουμε στο θέμα αυτό των αποθεμάτων. Άλλο σημείο, οι εγγυημένες τιμές όπως ισχύουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μεσαία επίπεδα και μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον για να μειώσουν τον κίνδυνο. Οι κίνδυνοι της εγγύησης, δεν μπορούν, οι ιδιωτικής εξασφάλισης δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την δημόσια πολιτική. Και η εφαρμογή ελάχιστων δικτύων ασφαλείας ε, είναι απαραίτητη ακόμη και αν το επίπεδό τους πρέπει να οριστεί σε χαμηλότερα επίπεδα, ώστε να μην ε, έχουμε στο μέλλον διόγκωση των αποθεμάτων. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κινδύνων. Η διαχείριση των κινδύνων είναι κάτι που απασχολεί την γεωργική πολιτική την τελευταία δεκαετία. Πάντως, η Γεωργή δεν είναι και πολύ ενημερωμένη στο θέμα αυτό όσο οικονομολόγοι τουλάχιστον για, όλα, για όλους τους μηχανισμούς που μπορεί να υπάρχουν. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, αυτό διαπιστώνω εγώ ως οικονομολόγος, μεγάλη διαφορά μεταξύ του φόβου που έχουμε για τους δυνάμει μηχανισμούς που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και για τον τρόπο που οι γεωργοί, ιδιαίτερα η εκτροφείς, οι κτηνοτρόφοι, είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους μηχανισμούς. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κινδύνων, ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης είναι η, η διατήρηση των δικτύων ασφαλείας και επίση ε, αρχή της προνοητικότητα στι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Στη Γαλλία νομίζω ότι επενδύονται πολλά κονδύλια στα γεωργικά εργαλεία. Κάτι που επιβαρύνει την ε, γεωργική οικονομία. Και οι δημοσιονομικές πολιτικές, οι φορολογικές πολιτικές είναι κατάλληλες για την προνοητική αποταμίευση που είναι η μεγαλύτερη εξασφάλιση και μεγαλύτερη εγγύηση για την θέση του Γεωργού ως προς τον μελλοντικό κίνδυνο. Στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι δείκτες διαχείρισης των κινδύνων να είναι πιο ελαστικοί από τους ισχύοντες. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να τους αξιοποιήσουμε. γιατί οι περιορισμοί για το πράσινο κουτί σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των, κινδύνων είναι, είναι πολύ περιορισμένοι. Επίσης θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και τις εμπειρίες των άλλων χωρών. Να ενθαρρύνουμε την επιμόρφωση των γεωργών για να μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα τους κινδύνους. Καλύτερα να ενθαρρύνουμε στα κράτη-μέλη μία μεταφορά των κονδυλίων από τον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ προς νέο μηχανισμό διαχείρισης των κινδύνων. Πολιτικά έχει εξαγγελθεί μια τέτοια πρόθεση, υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί. Απλώς τα ποσά που διατέθηκαν για το σημείο αυτό είναι πολύ συχνά σε σχέση με τις προσδοκίες και τις ανάγκες. Σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις για την αγρανάπαυση, να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ο μηχανισμός της αγρανάπαυσης είχε ένα ποσοστό που ε, προσαρμοζόταν κάθε χρόνο στις εξελίξεις των τιμών της αγοράς ετηρών. 5% ε, ήταν μια φορά, άλλη χρονιά ήταν 15%, άλλη χρονιά ήταν 10%. Καλή αυτή η διακύμαση του ποσοστού και θα έπρεπε να την ε, κρατήσουμε και για τις ποσοστώσεις. Γαλακτοκομικές ποσοστώσεις για μένα είναι από τα πιο σημαντικά ντοσιέ, ίσως επειδή μεγάλος. Οι γαλακτοκομικές ποσοστώσεις επικρίθηκαν κατά τη στιγμή της έγκρισής τους. Σήμερα οι γεωργοί επικρίνουν την πρόταση κατάργησής τους. Πάντως η μεγάλη δυσκολία που θα αντιμετωπίσουμε στην Ευρώπη είναι ότι έχουμε εφαρμόσει ε, τι γαλακτοκομικές ποσοστώσεις εδώ και 25 χρόνια, αλλά με διαφορετικό τρόπο μεταξύ των χωρών μελών. Τίποτα, ε, καμία σχέση δεν έχει η εφαρμογή των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων στη Δανία και στη Γαλλία, για παράδειγμα. Γιατί στη μία περίπτωση έχουμε αγοραία ποσοστό στην άλλη μία αγοραία. Ε, στη μία περίπτωση έχουμε διαχείριση αγορά και στην άλλη διοικητική διαχείριση. Καμία σχέση λοιπόν η διαχείριση που κάνει κάθε χώρα για τι γαλακτοκομικέ τη ποσοστώσεις. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτόματα όμως μια ενιαία θέση για τον τρόπο ρύθμισης. Γιατί για 25 χρόνια επιτρέπαμε στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ε, αποκλίνουσες πολιτικές. Οι γαλακτοκομικές ποσοστώσεις είχαν κάποια πλέον δημοσιονομικά, εδαφικά αλλά και κοινωνικά. Το ζήτημα που ανακύπτει τώρα είναι θα πρέπει να καταργηθούν αυτές οι, οι, οι ποσοστώσεις. Αυτή η ερώτηση είναι ρητορική γιατί έχει ήδη ληφθεί απόφαση θα πρέπει να αυξηθούν κατά 1% το χρόνο μεταξύ 2009 και 2013, ώστε να μπορέσουμε να τις καταργήσουμε κάποια στιγμή. Πολύ κακή αυτή η στρατηγική κατά τη γνώμη μου. Είναι κακή αυτή η στρατηγική γιατί θα πρέπει να προβλέψουμε περισσότερα μέσα για μια πιο ελαστική μετάβαση και λιγότερο αφιλεγόμενη για τους πολίτες. Μια ε, ελαστική μετάβαση από, από μια κρατική σε μια ιδιωτική ρυθμίση. και όσο θα απομακρύνεται το κράτος να υπάρχει δυνατότητα για μεγαλύτερη απορρίθμιση. Άλλωστε οι Ευρωπαίοι παραγωγοί δεν εξάντλησαν τις γαλακτοκομικές προσωστώσεις, έμειναν 5 δισεκατομμύρια λίτρα γάλακτος ανεκμετάλλευτα. Η, αύξη, η πρόταση αύξηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων ίσω δεν είναι η καλύτερη διέξοδος για να προετοιμάσουμε το 2015. Αν καταργηθούν όμω οι γαλακτοκομικές ποσοστώσει, ποια είναι η ακολουθητέα στρατηγική. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπήρξε βραχυπρόθεσμη ανάγκη κατάργηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων εξαιτία του ΠΟΕ. Η κατάργηση προτάθηκε για άλλου λόγου. Αν καταργηθούν αυτέ οι γαλακτοκομικέ ποσοστώσει, με τι θα αντικατασταθούν. Θα πρέπει να δεχτούμε την ιδέα ότι πρόκειται ε, για μια αδιαφορία του κράτους μετά από 25χρονη πρακτική. Δεν έχουμε πολλούς τομείς που να εφάρμοσαν τέτοια μηχανισμό. Αυτή όμως η απομάκρυση του, του, του κράτους θα πρέπει να γίνει σταδιαία, βαθμιαία και με εγγυήσεις προς τους παραγωγούς. Εγώ θα ήθελα να ενισχυθεί η σύναψη συμβάσεων με τον ιδιωτικό τομέα. Αλλά βαθμιαία, με μεταβατικό τρόπο. Και θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στις χώρες όπου έχουν περισσότερες επιχειρήσεις να κρατήσουν αυτή τη συναψύμβαση σε εθνικό επίπεδο με εθνικούς κανόνες που θα είναι αρκετά ακμαίοι, αρκετά ρωμαλαίοι, ώστε να ε, δώσουν μια ασφάλεια στους γεωργούς. Επίσης να μην ε, επισπευθούν τα πράγματα σε χώρε όπως η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή κάτω χώρε που υιοθέτησαν διαφορετική μέθοδο. Μπορούμε να δεχτούμε την ιδέα της σταδιακής απομάκρυση του κράτους ε, από την οικονομική ρύθμιση του γαλακτοκομικού κλάδου, αλλά ο τρόπος που θα γίνει κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικός. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι η γαλακτοκομική κρίση δεν σχετίζεται με την υπερπαραγωγή γάλακτος. Είναι μια διεθνή κρίση και θα είχαμε μια ακόμη πιο τραγική κατάσταση αν ε, οι γεωργοί είχαν σεβαστεί την δυνατότητά τους, δηλαδή να εξαντλήσουν τις ποσοστώσεις. Επίσης, ως προς τη ρύθμιση, θα ήθελα να πω κάτι για τις άμεσες πληρωμές. Στη Γαλλία τελικά θα δεχθούμε την αποσύνδεση όλων των ενισχύσεων. Εδώ το επίδομα στις προβατίνες το αποσυνδέσαμε. Η αποσύνδεση αρχίζει και γενικεύεται. Μάλιστα αυτό δεν είναι πρόβλημα για τις ορεινές περιοχές, γιατί δεν έχουν ούτως ή άλλως επιλογή. Το, το θέμα της επίδομα της σε Ελλάδας δημιουργεί πρόβλημα στις πολυκαλλιέργειες και στις εκτροφές, γιατί έτσι δίνουμε πλεονέκτημα στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Ε, σε ό,τι αφορά τις αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις, όπως είπε και ο κύριος Μπάκουελ, διανύουμε μία επικίνδυνη περίοδο και είναι επικίνδυνη για τον απλούστατο λόγο ότι οι αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις δίνονται άσχετα από τις τιμές της αγοράς. Αυτή ήταν η μεγάλη μας ευτυχία και χαρά. Όταν είχαμε εκτόξευση της τιμής των σιτηρών στα ύψη, είχαμε ταυτόχρονα και ακρίβεια το, του γάλακτος. Μερικέ φορέ οι αγορέ έχουν διαφορετική συμπεριφορά. Για φανταστείτε να είχαμε αύξηση τη τιμή των σιδηρών και μείωση τη τιμή του γάλακτο. Τότε θα είχαμε εκρηκτική κατάσταση στην Ήπεθρο. Οι αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις που έχουν πολλές αρετές, πολλά πλανεκτήματα, αυτή τη στιγμή ε, υποφέρουν. Γιατί αν είχαμε μια αντίστροφη ρευστότητα των τιμών, θα ήταν ε, απαράδεκτη η διατήρηση του συστήματος. Θα πρέπει λοιπόν να επαναπροσανατολίσουμε αυτό το σύστημα. Το γεγονός ότι έχουμε μια τέτοια ενίσχυση, ενιαία ενίσχυση ανά εκτάριο, ανά θα λύσει το πρόβλημα της νομοποίησης, γιατί όσο περισσότερα εκτάρια έχει κανένας, τόσο περισσότερη ενίσχυση το θέμα της νομοποίησης της αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης έγκυται στην μετατροπή, της, μετατροπή ενός τμήματός της προς μία νέα ε, ενίσχυση που θα λαμβάνει υπόψη και το περιβάλλον. Είμαι υπέρ μιας ενιαίας αποσυνδεδεμένης ελάχιστης ενίσχυσης για τους Γιώργους και πέραν τούτου προτιμώ καλύτερη σύνδεση της καταβολής των αποσυνδεμένων ισχύσεων με την πραγματικότητα των μη αγοραίων υπηρεσιών που προσφέρουν οι γεωργοί. Και έρχομαι και προς το συμπέρασμά μου. Για έναν οικονομολόγο είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κατάσταση να παρατηρεί ε, τη γεωργία και να κάνει όλες αυτές τις θεωρίες περί γεωργίας και μερικές ε, εκθέσεις που συντάσσουμε εμείς είναι τελείως ε, άχρηστες ή αδιάφορες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κρίμα, τέλος πάντων. Πάντως στη Γεωργία όλοι αντιμετωπίζουμε ε, προβλήματα, αλλά Θέλουμε να είμαστε πιο παραγωγικοί, καινοτόμοι, ανταγωνιστικοί, να παραμείνουμε στην αγορά και προσανατολισμένοι προς τους καταναλωτές. Όλοι συμφωνούμε ως προς αυτούς τους στόχους για τη γεωργία. Το θέμα είναι πώς θα υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει στην Ευρώπη να εφαρμόσουμε μια ε, λιγότερο ευρωπαϊκή πολιτική. Η συγχρηματοδότηση έχει ένα πλεονέκτημα. Είναι ότι ε, εμπλέκει και τα κράτη στην ευθύνη της κατανομής των ενισχύσεων δεν θα πρέπει να απομακρυνθούμε από την ε, κοινοτική ιδέα. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Επίσης θέλουμε μια κοινή γεωργική πολιτική που θα είναι συμβατή με την ε, γεωργική ανάπτυξη και στις αφρικανικές χώρες, όπου εκεί η δημογραφική ανάπτυξη είναι τέτοια που τους υποχρεώνει να αναπτύξουν μόνοι τους τη γεωργία τους. Επίσης θέλουμε μια πιο δίκαιη κοινή γεωργική πολιτική. Γιατί ο κόσμος ε, ε, έχει χάσει την ανθρωπιά του. Μιλούσαμε πριν από 10 χρόνια για το ανώτατο όριο των ενισχύσεων. Όχι αναγιορική εκμετάλλευση. Είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Το ξέρουμε 15 χρόνια και. Αλλά ανά απασχόληση, αναθέση απασχόλησης. Ακόμη και με την επικουρικότητα μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα τέτοιο ανώτατο όριο. Δεν νομίζω ότι είναι επαναστατική μια τέτοια ιδέα το 2009, παρόλο που όταν πρωτοπαρουσιάστηκε είχε ένα τέτοιο χαρακτήρα. Είμαι υπέρ μιας ρυθμισμένης γεωργίας με τη διατήρηση κάποιων δικτύων ασφαλείας. Χρειαζόμαστε αυτά τα δικτύα ασφαλείας, τις εγγυημένες τιμές, γιατί προστατεύουν τους γεωργούς και τους δίνουν την αίσθηση ότι το κράτος ενδιαφέρεται έστω και λίγο για την κατάσταση των τιμών των προϊόντων τους. Επίσης, η σύναψη των συμβάσεων αντικαθιστά την πολιτική γαλακτοκομικών ποσοστώσεων ή η κατανομή της προστιθέμενης αξίας, η κατανομή του κέρδους. Και αυτό είναι πολύ περίπλοκο θέμα που συνδέεται άμεσα με τον ε, τρόπο που θα σχεδιάσουμε το μέλλον της ΚΑΠ. 30 δισεκατομμύρια ευρώ αποσυνδεμένων ενισχύσεων που δίνονται στους γεωργούς με βάση κυρίως ε, την ιστορική αναφορά και όχι με βάση την παρούσα οικονομική τους κατάσταση ούτε με βάση των μη αγοραίων αγαθών που προσφέρουν ή τουλάχιστον ε, ελάχιστα. Ούτε ε, σε σχέση με το, προσωπικό τους όραμα. Νομίζω ότι μια τέτοια πολιτική που στηρίζεται στις ιστορικές αναφορές θα πρέπει να αλλάξει αμέσως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Σατελιέ για αυτή την ε, πολύ σημαντική συνεισφορά. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπάκουερ, φυσικά τον προηγούμενο ομιλητή. Ξεκινάμε ένα πρώτο γύρο παρατηρήσεων. Θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα και στην Επίτροπο να ακούσει τις πρώτες αντιδράσεις των μελών της Επιτροπής μας. Ε, τώρα ξεκινάμε με τους συντονιστές των ομάδων. Ο κ. Άλμπερτες, πρώτος και καλύτερο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την διοργάνωση του εργαστηρίου αυτού. Νομίζω ότι ακούσαμε διάφορα επιχειρήματα και θα δεν θα ήθελα και εγώ να κάνω παρουσίαση, απλά θα ήθελα να σχολιάσω. Καταρχάς, ε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας ε, μιλάτε για αυτό το ανεπίσημο έγγραφο. Το διάβασα το ανεπίσημο έγγραφο και πρέπει να σας πω ότι έχει προηγηθεί πολλή δουλειά. Αν λοιπόν έχει γίνει τέτοια δουλειά από υπαλλήλου. Μήπως θα έπρεπε να κοιτάξουμε γιατί απασχολούνται τόσα άτομα. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι κάθισαν και ασχολήθηκαν τόσοι άνθρωποι με αυτό το έγγραφο για το θέμα το οποίο συζητήθηκε σήμερα για την ΚΑΠ μετά το 2013. Ακούστηκαν επικριτικές, επικριτικά σχόλια για τις πληρωμές. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να τα κοιτάξουμε και με κάποιο σχετικό πνεύμα. Το 1970 ήταν ακόμα στο 87%. Τώρα είμαστε στο 76%. Το 2013 θα είμαστε γύρω στο 36%. Εξακολουθεί να είναι υψηλό το ποσοστό. Μιλάμε όμως για το 5% του πληθυσμού της Ευρώπης. Θα πρέπει να το σχετικοποιήσουμε όμως το ποσοστό αυτό. Αν ε, όλες οι πολιτικές ρυθμίζονται από τις Βρυξέλλες, Μιλάμε για το 3% το οποίο δαπανάται για το 5% του πληθυσμού. Ασκούμε δηλαδή πολιτική για 500 εκατομμύρια καταναλωτές στην Ευρώπη. Αν μιλάμε και ας κάνουμε μια στογγυλοποίηση ε, του ποσού. Αν πούμε για 500 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη θα πανώνται 50 δισεκατομμύρια. Μιλάμε δηλαδή για 100 ε, ευρώ ανά κάτοικο το έτος και μιλάμε για την διατροφική ασφάλεια, για τη φροντίδα του περιβάλλοντος. Μιλάμε για την πιο ε, φτηνή ασφάλεια ζωής στην Ευρώπη. Και τι θέλουμε για την περίοδο μετά το 2013 μια εύλογη κατανομή των δαπανών αυτών. Θα πρέπει να γίνουν λοιπόν σωστές προτάσεις, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να τηρούνται σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, για παράδειγμα, με το 2013, ακόμα πιο αυστηρά πρότυπα. στο δεύτερο πυλώνα ξεκινάμε για τις ε, μειονεκτικές περιοχές και εξισορρόπηση των δαπανών. Θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια εξισορρόπηση, γιατί δεν θα καταφέρουμε σε εποχές που είναι ανοιχτά τα σύνορα να περιορίσουμε τις αγοράες. Θα πρέπει όμως να δώσουμε τις ευκαιρίες τις κατάλληλες προς τους ε, αγρότες και κυρία Επίτροπε. Είπατε ότι δεν θα συμμετέχετε στην επόμενη Επιτροπή. Κάνατε μία σωστή παρατηρήση και θα ήθελα να την υποστηρίξω. Πρέπει η διατροφική ασφάλεια να διασφαλιστεί και για το μέλλον για 50 εκατομμύρια άτομα. Δεν μπορούμε λοιπόν βάσει κάποιων εξελίξεων στην παγκόσμια χώρα να βγούμε και να πούμε ότι α, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε με τις τιμές αυτές. Γιατί υπήρχαν ε, οικονομολόγοι που βγήκαν πριν από 5-6 χρόνια και είπαν γιατί θέλουμε βιομηχανία χάλιβα στη Γερμανία, αφού μπορούμε να εισάγουμε χάλιβα από τη Βραζιλία. Και τι έγινε, στη συνέχεια τετραπλασιάστηκαν τετραπλασιάστηκε η φορολογία. Για φανταστείτε να γίνει κάτι τέτοιο, να τετραπλασιαστούν οι τιμές για την, τα τρόφιμα για, 500 εκατομμύρια ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι απαραίτητη η πολιτική αυτή και για την περίοδο μετά το 2013. Πρέπει να ζητήσουμε μία οδό για το πώς θα διαμορφωθεί από το 2014 και μετά η πολιτική αυτή. Ευχαριστώ, Άλμπερτ. Ε, Λουίς Κάπουλα Σάντος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου Γεωργίας, την Επίτροπο και τους εμπειρογνώμονες που μας έδωσαν την έγκριτη τους γνώμη. Θα ήθελα να πω κάτι προς την Επίτροπο Officer Bull, Bell. Κατά πάσα πιθανότητα είναι η τελευταία φορά που έρχεστε στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα και προσωπικά, αλλά και εκ μέρους πολιτικής μου ομάδας, να σας εκφράσω την απεριόριστη εκτίμηση και αναγνώριση που τρέφουμε προς το πρόσωπό σας. Και θα σας εξομολογηθώ και κάτι προς αυτό το κατάμεστο κροατήριο. Ε, ως υπουργό ε, μια μεγάλη χειρονομία αλληλεγγύης. Και για να επιλύσετε ένα πρόβλημα της πατρίδας μου, της Πορτογαλίας, θυσιάσατε ένα τμήμα του πολιτικού σας γοήτρου στην ε, Δανία. Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσω αυτή την αλληλέγγυα χειρονομία σας. Γι' αυτό έχουμε πολύ καλές εντυπώσεις και αναμνήσεις ε, από σας. Έχετε πάρα πολλές αρετές, αλλά ένα μικρό μειονέκτημα έχετε, είστε υπερβολικά φιλελεύθεροι, αλλά χρόνο έχετε, μπορεί να το διορθώσετε στην ε, μελλοντική σας σταδιοδρομία. Πάντως, επαναλαμβάνω, τρέφουμε ιδιαίτερη εκτίμηση προς το πρόσωπό σας και χαίρομαι για τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια για την συγκεκριμένη εντολή και την ε, τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα ξαναγράψουμε ένα τμήμα της ε, ευρωπαϊκής ιστορίας. Γιατί η κοινή γεωργική πολιτική και το μέλλον της ΚΑΠ είναι άμεσα συνειφασμένα με το μέλλον του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Θα πρετανεύσουν ε, τα εθνικά συμφέροντα και οι εθνικοί εγωισμοί ή θα θα θυσιάσουμε αυτά στο όνομα μιας κοινή γεωργικής πολιτικής. Η σημερινή ΚΑΠ είναι μια ΚΑΠ που σχεδιάστηκε αρχικά για 6 χώρες, μετά για 9, για 10, για 12 και μετά για 15 χώρες. Ήταν λοιπόν μια γεωργική πολιτική που στην πρόσφατη ιστορία της περνούσε από αλλαγή σε αλλαγή και από προσαρμογή σε προσαρμογή. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι φτάσαμε σε μια φάση όπου θα σταματήσουν οι διευρύνσει. Και το 2013 θα τελειώσει και η σταδιακή ένταξη των νέων χωρών. Οπότε δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη χάραξη μια γνήσια πολιτική για 27, 28, 29 χώρε. και θα δούμε αν πραγματικά είμαστε ικανοί να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία. Ξέρω ότι δεν έχω χρόνο, γι' αυτό δεν θα μακρηγορήσω, αλλά θα ήθελα να σας βάλω μία πρόκληση. Καταρχήν για τους εμπειρογνώμονες. Οι εξηγήσει σας επιβεβαίωσαν ε, τη θέση μου και αυτό που υποστηρίζω εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί από το 1992 έχουμε ένα μοντέλο που ήταν προκαθορισμένο και είχε ε, προβλέψιμη πορεία. Είναι αδύνατο να την παρεκκλίνουμε. Από τη στιγμή που ξεκινάει ένα πύραυλο, δεν μπορούμε να παρεκτρέψουμε την πορεία του, ούτε να τη διορθώσουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με την ΚΑΠ, που η πορεία τη είναι προδιαγραμμένη. Η ερώτηση που έχω προς τους εμπειρογνώμονες είναι η εξή. Παρόλο που ήταν σαφέστατες οι παρεμβάσεις, ιδιαίτερα του κυρίου Μπάκουελ, έχει νόημα μετά το 2013 να κρατήσουμε τους δύο πυλώνες. Κατά τη γνώμη μου όχι. Γιατί από αυτά που ακούσαμε διαπιστώσαμε ότι στο μέλλον δεν θα έχει νόημα να έχουμε δύο πυλώνες στην γεωργική πολιτική. Αυτό το υποστήριζα εδώ και χρόνια και θα ήθελα να μου το σχολιάσετε. Η πρόκληση λοιπόν που έχουμε και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο είναι αν θα έχουμε την πολιτική τόλμη στο μέλλον και αν θα δείξουμε το θάρρος για να διαμορφώσουμε μια κοινή γεωρική πολιτική που δεν θα είναι μόνο μια απλή συζήτηση γύρω από τα εθνικά κονδύλια, αλλά θα είναι μια γνήσια κοινή πολιτική, όπως είπε και η Επίτροπος, που θα δώσει στην Ευρώπη συνοχή, αλληλεγγύη και θα προσπίσει το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας και της Υπέθρου που αν δεν υπάρχει τέτοια πολιτική θα είναι αβέβαιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Λουίς, ευχαριστώ για την πολύ σημαντική έτσι και γεμάτο, γεμάτη πάθος παρέμβασή σου. Ε, η Επίτροπος μπορεί να παραμείνει, θα το λόγο στον George Λάιον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου όλους ε, τους ομιλητές και κυρίως ε, τον πρόεδρο, τον του Συμβουλίου και τη Μαριάν Φίσοκ Μπόλ, η οποία ακόμα μια φορά έκανε μια πολύ στενάρη έτσι παρουσίαση. Χαίρομαι ε, που άκουσα ότι αυτό το έγγραφο δεν ε, υπάρχει και μπαίνει στα σκουπίδια, όπως και άλλοι χάρηκαν. Θα ήθελα να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο δεν υπογραμμίστηκε μέχρι στιγμή στη συζήτησή μας αρκετά. Δέχομαι την ανάγκη να προσφέρει δημόσια αγαθά η ΚΑΠ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να στηρίζεται και στην αποδοχή του κόσμου, ε, στη διαχείριση της γης, ε, ε, πρότυπα ευημερίας, περιβάλλον, καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και αυτό θα πρέπει να ενταχθεί στους μελλοντικούς στόχους της ΚΑΠ. Ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε αγγίξει είναι μια ανταγωνιστική γεωργική, γεωργικός τομέας στην Ευρώπη. Ε, βλέπουμε άλλε χώρε όπω οι Ηνωμένε οι οποίες έχουν συστήματα υποστήριξης που επεκτείνονται με επιθετικό τρόπο. Ε, με το πρόσφατο νομοσχέδιο για τη Γεωργία του 2008 ενίσχυσαν το σύστημα των πληρωμών, όπως ονομάζεται, και ενίσχυσαν επίσης και το σύστημα ασφάλισης εναντίον κινδύνων. Ε, ο κλάδος της, τον είπα, θα υποστηριχθεί και από κυβερνητικές παρεμβάσεις σε περίπτωση κρίσεων. Ε, ούτως ώστε να μπορεί να αναπτύσσεται και να γίνεται πιο ανταγωνιστικό στο μέλλον. Επομένως, από ό,τι φαίνεται, οι δεσμεύσεις μας ε, στον ΠΟΕ είναι τέτοιες ε, που μας θέτουν σε καλύτερη θέση αυτή τη στιγμή έναντι των ΗΠΑ. Το θέμα είναι, αναπτύσσουμε μια πολιτική η οποία θα έχει μια μειωμένη ε, παραγωγικότητα, μειωμένη δηλαδή ε, παραγωγικότητα η γεωργία της ε, Ευρώπης. Αυτό σημαίνει πιο ρευστή και ασταθή κατάσταση παραγωγής και τοπικής παροχής προϊόντων αν ε, αρχίσει να φθήνει η γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλοι θα μπουν για να καλύψουν το κενό με τις εξαγωγές κτλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ΚΑΠ ε, είναι ανταγωνιστική και γεμίζει τα στομάχια των Ευρωπαίων πολιτών. Δίνει προϊόντα στους καταναλωτές τα οποία χρειάζονται. Θα πρέπει μια πολιτική δηλαδή να ικανοποιεί αυτό που θέλει το κοινό να είναι, ανταγωνιστική, να είναι ανταγωνιστικός κλάδος, που θα μπορεί επίσης να ανταγωνιστεί και σε διεθνές επίπεδο. Ε, επειδή έχουμε ανώτατο όριο στον προπολογισμό, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν και οι Αμερικανοί γεωργοί το ίδιο πρόβλημα. Ε, δεν λέει καθόλου ο Αμερικανικός προπολογισμό. Όταν φτάσετε σε αυτό το ανώτατο επίπεδο, τέρμα υποστήριξη, Οποιαδήποτε και αν είναι τα, οι ανάγκες ε, των Αμερικανών γεωργών σε περίπτωση κρίση, ε, ο προπολογισμό υπάρχει εκεί για να το στηρίξει. Χρειαζόμαστε και εμείς ανταγωνιστική γεωργία και ανησυχώ ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που μας απασχολεί είναι ε, το θέμα της περικοπής του προπολογισμού. Νομίζω ότι πρέπει και εμείς να είμαστε επιθετικοί και θα πρέπει να υποστηρίξουμε μια βιώσιμη ανταγωνιστική γεωργία και που δίνει α, υπηρεσίες και αγαθά στους, στο κοινό ακριβώς αυτά που περιμένει να δει. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, George. Τελειώνουμε τον ε, κύκλο των παρεμβάσεων των ε, συντονιστών με τον Μάρτιν Χόστιν και συνεχεία θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο ο Εσκύλ είπε ότι δεν θέλει να παρέμβει. Ο Μάρτιν λοιπόν έχει το λόγο. Νομίζω ότι, νομίζω ότι πρόκειται για μια συζήτηση πολύ επικοδομητική και νομίζω ότι μιλάμε για μη επίσημα έγγραφα τα οποία καταλήγουν στο καλάδι των χρήστων. Δεν πρόκειται για σύμπτωση όμως, γιατί αυτή είναι η πολιτική που θέλουμε να κάνουμε καταρχάς θα πρέπει να, να συμφωνήσουμε επί των στόχων και μετά να δούμε σε τι χρηματοοικονομικό πλαίσιο θα πρέπει να τεθούν. Όχι αντίστροφα. Στην όλη συζήτηση μου έκανε εντύπωση ότι λείπαν δύο στοιχεία. Καταρχάς, ότι Μιλάμε για ανθρώπους για θέσεις εργασίας. Και για σημαντικούς αριθμούς. Θα πρέπει να το λαμβάνουμε αυτό υπόψη όταν μιλάμε για την μεταρρύθμιση του κλάδου. Κάτι που είπατε κυρία Φίσερ Μπέλ. Είπατε ότι αδίκως σας ε, χαρακτηρίζουν πολύ φιλελεύθεροι. Είσαστε όμως πάρα πολύ φιλελεύθεροι στην ε, γεωργική πολιτική. Είπατε ότι θα πρέπει να προσανατολιστούμε στις ε, παγκόσμιες αγορές. Νομίζω ότι αυτή η πολιτική, όπως μας έδειξαν τα τελευταία δύο χρόνια, δεν μπορεί να συντηρηθεί. Θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια σωστή διαχείριση. Και όταν λέμε ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των γεωργών, χρειάζεται και μία συζήτηση για το πώς θα μπορούμε να κατευθύνουμε τη ζήτηση, πώς μπορούμε να τους δώσουμε στους αγρότες μέσα για να καθορίσουν αυτή το μέλλον τους. Όλα αυτά είναι σημαντικά, για παράδειγμα και σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις. Σε ένα πράγμα συμφωνούμε, ότι στις μερατικές πληρωμές θα παίξουν σημαντικό ρόλο οι περιβαλλοντικές διαστάσεις. Το 9% που ακούσαμε για τις εκπομπές του άνθρακα που προέρχεται από τη γεωργία δεν νομίζω ότι είναι σωστό, γιατί πρέπει να συνυπολογίσουμε και τις δευτερογενείς ε, επιπτώσεις. Και τι προστίθεται και από τη Βραζιλία, από τη ΣΥΠΑ. Και όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν λοιπόν στον ενεργειακό ισολογισμό και θα πρέπει να το σκεφτούμε καλά. Γι' αυτό δεν πιστεύω το επιχείρημά σας για αύξηση κατά 45%. Δεν ξέρω αν εννοούσατε τη δική μας γεωργία αποκλειστικά για να θρέψουμε τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να θρέψουμε τον ε, κόσμο με χείριο κρέας μόνο. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον τρίτο κόσμο. Όχι μόνο να λαμβάνουμε υπόψη ναι, τη δική μας ε, κοινωνία, τη δική μας κοινωνία που τρέφεται τόσο πολύ με πρωτεΐνες για παράδειγμα. Την όλη συζήτηση για τους πυλώνες θα πρέπει να παρακολουθήσουμε την όλη κατεύθυνση. Εμείς οι πράσινοι λέμε ότι θέλουμε την ε, πτυχή του δεύτερου πυλώνα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της πέτρου, για παράδειγμα. Θέλουμε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή και στις πληρωμές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μια τεράστια ανισορροπία σε ό,τι αφορά τους αποδέκτες, δηλαδή όσοι εποφελούνται από τον πρώτο πυλώνα έχουν τις πιο μεγάλες επιφάνειες και αυτοί που λαμβάνουν πιο λίγα, δηλαδή οι μικρές επιχειρήσεις. Πρέπει κάθε φορά να ε, δικαιολογούν τις πληρωμές αυτές. Μαριάν Φίσορμπόλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Παύλο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Καταρχάς, για αυτό το non-paper. Δεν το έφτιαξε η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, έτσι, το λέω ξεκάθαρα. Και δεν πέρασε μέσα από την από τα κλασικά κανάλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο γεω... γεωργικός προπολογισμό θα παραμείνει ακέραιος στο μέλλον. Θα πρέπει να προετοιμαστείτε ε, για μεγάλα σοκ. Ε, και πολλοί καρχαρίες θα θελήσουν να αρπάξουν ένα κομμάτι από το γεωργικό προπολογισμό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ισχυρά επιχειρήματα για να εξηγήσουμε γιατί χρειαζόμαστε στο μέλλον την κοινή γεωργική πολιτική. Θα γίνει λοιπόν αυτή η συζήτηση αλλά όταν ε, θα υπάρξει το νέο κείμενο, το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει, θα έχει περάσει μέσα από τα σωστά κανάλια και θα έχει εγκριθεί από το Σώμα των Επιτρόπων πριν ε, δημοσιευθεί. Δες. Συμφωνούμε μαζί. Συμφωνούμε ότι έχουμε διάφορα τεράστια νούμερα για το μερίδιο της ΚΑΠΑ στον προπολογισμό και που συνδέονται και που συνδέεται με το ΑΕΠ των κάτων μελών. Εδώ το 0,43% είναι αυτό που παίρνει η Γεωργία σε σχέση με το κοινοτικό ΑΕΠ. Αν το συγκρίνετε με το προπολογισμό της, για την άμυνα, ε, είναι τέσσερι φορέ μεγαλύτερη. Επομένω, αυτή η ασφάλεια που μα δίνει η Γεωργία δεν, τόσο, δεν την πληρώνουμε πολύ ακριβά. Θα πρέπει αυτό το νούμερο το 0,43% να το πούμε στον κόσμο. Ξέρετε την άποψή μου για την ανάπτυξη τη υπαίθρου. Νομίζω ότι στο μέλλον θα πρέπει να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στι πολιτικέ μα η ανάπτυξη της υπαίθρου. Χρειαζόμαστε να εστιάσουμε πιο συγκεκριμένα ε, στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η, ανα... η ανάπτυξη της υπαίθρου, ε, κλιματικές ε, αλλαγές, ε, νερό και βιοπικιλότητα, καθώς και ενέργεια. Τέσσερις προκλήσεις. Φυσικά από, αυτές τις τέσσερις, από αυτά τα τέσσερα στοιχεία μπορούν να διαλέξουν πού θέλουν να εστιάσουν τα κρατη γιατί δεν συμφωνούν ποτέ όλοι. Θα ήθελα η πολιτική αυτή να παίξει τον ρόλο του καρότου, ούτως ώστε οι γεωργοί να αισθάνονται ότι ε, έχει νόημα να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέτρα και να δώσουν μια έτσι, ποικιλόμορφη γεωργία. Αν ε, όμως αυξήσουμε τα κονδύλια για, τις, ε, για την ανάπτυξη υπαίθρου, θα πρέπει να μειώσουμε τις ε, άμεσες ε, ενισχύσεις. στο μέλλον δεν νομίζω θα έχουμε το άρθρο 66. Όταν αν δημιουργήσουμε νέες πολιτικές, τότε αυτά τα εργαλεία θα μείνουν έξω. προφανώς γι' αυτό θα αναπτύξουμε, αν αναπτύξουμε νέα στοιχεία. Ο Καπούλα Σάντος. Στο μέλλον, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι τεράστιος. Πολύ κρίσιμος, πολύ σημαντικός. Αυτό μας θα απαιτήσει από εσά να δείξετε γενναιότητα και συχνά να λάβετε τις άρεστες αποφάσεις. Τότε θα μπορείτε να κρυφτείτε ότι η Επιτροπή είναι κακή, ότι η Επιτροπή αποφασίζει μαζί με το Συμβούλιο. Και εσείς θα πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη που σας αναλογεί. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Ε, εγώ θα σας έχω στο μάτι πάντα. Θα βλέπω, θα σας παρακολουθώ πώς θα τα καταφέρετε να ξεφύγετε από τις δυσκολίες, να τις αντιμετωπίσετε τις ε, δυσκολίες για τα δημόσια αγαθά. Συμφωνούμε για αυτό το θέμα. Δεν νομίζω όμως ότι είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε και να εντοπίσουμε τις μελλοντικέ πολιτικές, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό. Για τον ΠΟΕ, κύριε Λάιον, για μένα είναι σαφές ότι ένας από τους λόγους για την ύπαρξη των συμφωνιών ΠΟΕ είναι γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να καναλιζάρουμε και να υπάρξει εσωτερική υποστήριξη. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό το νομοσχέδιο το αμερικανικό ε, προκαλεί στρεβλό στον ανταγωνισμό, γιατί δεν υπάρχει... Είναι απεριόριστα τα κονδύλια που μπορούν να δοθούν. Σε αυτή τη φάση δεν είμαι πολύ αισιόδοξη, αλλά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το θέμα. Φυσικά υποστηρίζω τις διμερείς εμπορικές ε, συμφωνίες, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσετε να ρυθμίσετε τέτοια γεωργικά θέματα μέσω διμερών συμφωνιών. Επομένω, το πολυμερέ επίπεδο είναι το καλύτερο. Επίση, κάποιοι άλλοι θα έρθουν και θα καλύψουν τα κενά αν εμεί δεν παράγουμε στην Ευρώπη. Σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βασιστούμε στα δυνατά μα χαρτιά, γιατί έχουμε μια πολύ καλή φήμη για ποιοτική παραγωγή. Και νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη φήμη όταν ε, ανακάμψουμε από τη χρηματοπιστωτική κρίση και να στραφούμε ειδικά προς τις ασιατικές αγορές. Δεν θεωρώ ότι η Ευρώπη πρέπει να παράγει μόνο για τους Ευρωπαίους. Ούτως ή άλλως σήμερα είμαστε και μεγαλύτερος ε, εισαγωγέας και εξαγωγέας γεωργικών αγαθών και νομίζω ότι έτσι θα συνεχιστεί. Παρά το γεγονός ότι όταν μεταφέρεται αγαθά ανά τον κόσμο, εκπέμπεται ε, αέρια του θερμοκηπίου. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά υπάρχουν κάποιοι τρόποι για να μειώσουμε τις εκπομπές μας. Κύριε Χάσλιν, ναι, είμαι φιλελεύθερη και είμαι περήφανη που είμαι. Αλλά αυτοί που λένε ότι είμαι υπερβολικά φιλελεύθερη, ε, φανατικά φιλελεύθερη, σφάλουν. Νομίζω ότι αν δεν έχεις το κουράγιο να λάβεις αυτές τις σκληρές και δυσάρεστες αποφάσεις και να ε, αλλάξει την ΚΑΠ, δεν νομίζω ότι ε, ετοιμάζουμε την ε, γεωργική πολιτική του μέλλοντος. Αν κάποια στιγμή δεν, πιέσου, δεν δεχτείς πιέσεις ε, ως γεωργός, γιατί να αλλάξεις. Μια χαρά είναι έτσι τα πράγματα. Κι όμως πρέπει καμιά φορά να στραφείς αλλού. Θα πρέπει να κάνεις αλλαγές. Εμείς θα πρέπει να έχουμε το πολιτικό θάρρος να κάνουμε αυτές τις πιέσεις. Φυσικά θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι κάνουμε το σωστό. Είμαι σίγουρη ότι η Ευρωπαϊκή Γεωργία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις αυτού του πιο παγκοσμιοποιημένου εμπορικού μοντέλου ε, και για τα γεωργικά προϊόντα. Γιατί έχουμε κάποια του στα χέρια μας για τις εκπομπές των ε, αερίων του θερμοκηπίου. Είναι 9%. Αλλά αν ε, μετρήσουμε και όλες τις ε, εισαγωγές, ναι, πρέπει να κρατήσουμε την παραγωγή κρέατος στην ε, Ευρώπη. Ε, αν λάβουμε υπόψη μας τα, τους κόκκους σόγιας κτλ. Ε, εκπέμπουμε όταν εισάγουμε και εκπέμπουμε όταν εξάγουμε. Θα πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή μας ε, μέχρι το 2050 κατά 70 με 100%. Έχουμε δυνατότητες αύξησης παραγωγής μας πρέπει όμως να, να το κάνουμε ε, να Παράλληλα με την αύξηση αυτή να βοηθήσουμε και τι αναπτυσσόμενε χώρε για να αυξήσουν την παραγωγή του. Γι' αυτό πέρυσι δώσαμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ για να αγοράσουμε σπόρου και λοιπάσματα για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Ε, το έχω πει αυτό. Αν τα δώσουμε αυτά, αν δώσουμε αυτά εργαλεία στι ε, γυναίκε, κάτι ε, θα συμβεί, κάτι θα κουνηθεί. Αν τα δώσει στους άντρε, τίποτα δεν γίνεται. Δεν το λέω για πλάκα. Οι άντρες κάθονται, αράζουν πίσω στις καρέκλες τους. Στο, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, στο ΦΑΟ, στη Ρώμη, στη συνάντηση αυτή θα πρέπει να βρούμε λύσει. Γιατί σήμερα ένα εκατομμύριο άνθρωποι παγκόσμια ημοκτονούν. Ο, οι στόχοι της χιλιετίας έλεγαν ότι θα πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των λιμοκτονούντων από 800.000 σε 400.000. Αυτό έχει αποτύχει. Αυτός ο στόχος δεν έχει υλοποιηθεί. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, τουλάχιστον για να θρέψουν τον εαυτό τους. Ευχαριστώ Παύλο. Ευχαριστώ Μαριάν. Και τώρα ένα-δύο λεπτά διαλύματος για να χαιρετήσω τη Μαριάν η οποία θα φύγει και να χαιρετήσω και τον Εσκύλ Και βεβαίως, για να τονίσω, νομίζω ότι εκφράζω έτσι το δημόσιο αίσθημα, την ευγνωμοσύνη μας για τη δουλειά που έκανε η Μαριάν αυτή την θητεία. Ε, νομίζω εκτιμούμε αυτή την προσπάθειά της. Ο καθένας βέβαια υπερασπίστηκε τις ιδέες του, αλλά νομίζω η Μαριάν πάνω απ' όλα υπερασπίστηκε την Ευρωπαϊκή Γεωργία, ε, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική η ευρωπαϊκή πολιτική. Ευχαριστώ όλους. Ένα-δύο λεπτά διάλειμμα για να χαιρετήσω τη Μαριάν. Would you then allow me just Οπότε επιτρέψτε μου με τη σειρά μου να πω δύο λόγια. Δεν ξέρω αν θα είναι η τελευταία φορά. Δεν ξέρω αν ε, θα με διώξουν από το αξιωμά μου. Μπορείτε να τα ξαναπούμε. Πάντως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Με κάποιους δεν, σας... δεν είμαστε γνωστοί, έτσι παλιοί γνωστοί, αλλά με κάποιους είμαστε γνώριμοι τα τελευταία πέντε χρόνια. Και πραγματικά ήταν μεγάλη χαρά να έρχομαι εδώ στο Κοινοβούλιο, να συζητάω μαζί σας, να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Δεν ήταν πάντα εύκολη δουλειά, γιατί δεν συμφωνούσαμε πάντα. Αλλά η χαρά να συνεργαζόμαστε ήταν μεγάλη. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, θα σας έχω στο μάτι. Ε, πώς θα διαχειριστείτε την νέα σας εξουσία. Ελπίζω να τα καταφέρετε. Αλλά χρειάζεται να, κάνετε, να πάρετε δύσκολες αποφάσεις. αλλά είμαι σίγουρη θα το κάνετε για το καλό της, του γεωργικού τομέα. Που γεωργία δεν σημαίνει στο τέλος μόνο προστασία, σημαίνει μερικές φορές και άνοιγμα της γεωργίας στις νέες προκλήσεις. Καλή τύχη. Bene, riprendiamo. Πολύ ωραία. Ξαναρχίζουμε. Τη εργασία μα. Τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον καθηγητή Εντουάρντο Ράμος από το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβας. Έχετε το λόγο για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής ε, ανάπτυξης της υπαίθρου. Θα χρειαστεί ένα-δύο λεπτά ε, για να χαιρετήσει τους εισηγητές η Μαριάν πριν βγει. Περιμένουμε. Tranquillo. He's talking with the Ramos. Maybe more. Maria.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 Okay. Eduardo Ramos is here. Is ready. Ο κύριος Ράμος είναι εδώ. Είναι έτοιμος. Prego. La parola Eduardo Ramos, l'Università di Porto. Ε, το λόγο, κύριε Ράμος. Muchas gracias, señor presidente. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης για την ευκαιρία που μου δίνει να συμβάλλω κι εγώ με τη μελέτη μιας ομάδας καθηγητών του Τμήματος οικονομίας, Αγροτικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου της Κόρδοβα. Δεν είναι οι προσωπικές μου απόψεις που σας μεταφέρω, αλλά σύσσωμες της ομάδας εργασίας στην οποία ανήκω. Θα ήθελα, πριν περάσω στην παρέμβασή μου, να σας προειδοποιήσω ότι όταν μιλώ για τον πρώτο πυλώνα, ενώ τις ε, άμεσες ενισχύσεις. Γιατί παρόλο που θα μιλήσω για τη μεταρρύθμιση πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, που ανήκει στο δεύτερο πυλώνα, θα κάνω και κάποιες συνήξεις για τον πρώτο πυλώνα και ιδιαίτερα για τις άμεσες ενισχύσεις, που είναι και το μεγαλύτερο τμήμα το πιο αντιπροσωπευτικό τμήμα του πρώτου πυλώνα. Εργάζομαι εδώ και περίπου 30 χρόνια σε θέματα αγροτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα και κάθε φορά που λάμβανε χώρα μια μεταρρύθμιση της ε, γεωργικής πολιτικής διαπίστωνα ότι πολλοί γεωργοί ήταν κατά της μεταρρύθμισης. Και μάλιστα στην Ισπανία που έχουμε ακραίες θέσεις η εμπειρία μας έδειξε ότι ποτέ δεν είχαν και ποτέ δεν δικαίωσε η πράξη τους γεωργούς. Δεν δικαίωσε τις αντιδράσεις τους. Αυτή τη φορά όμως, ε, επειδή είναι διαφορετικά τα πράγματα και ο φόβος τους ε, δικαιολογείται, αυτή τη φορά δικαιώνονται οι αντιρρήσεις των γεωργών γιατί από άμεσε έρευνε που κάναμε στι γεωργικέ εκμεταλλεύσει, γιατί είναι διτό ο χαρακτήρα τη οικονομία. Μερικέ φορέ μιλούμε για την αδύναμη γεωργία και την ανταγωνιστική γεωργία. Αλλά πρόκειται για ένα δίπτυχο. Συνυπάρχουν αυτέ οι δύο μορφέ γεωργία, και η αδύναμη και η εύρωστη. Και δεν μπορούμε να μιλούμε για τη μία και να κάνουμε σαν να μην υπάρχει άλλη. Η πιο ανταγωνιστική γεωργία, που είναι η, ο τομέας των απορροκυπευτικών της Μεσογείου, που είναι σχετικά αριθμιστος τομέας, ε, και δεν λαμβάνει πολλές ενισχύσει. Ε, διανύει αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί παρόλο που έκαναν πολλές επενδύσεις στο κλάδο, είχαν πολύ αυστηρέ προσαρμογές, τους έπιασε και κρίση και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τραπεζική χρηματοδότηση για να αντιμετωπίσουν αυτή την αρνητική συγκυρία και οι άνθρωποι τα έχουν χαμένα, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Συμφωνώ με τον Γάλλο οικονομολόγο ότι η αβεβαιότητα είναι ο χειρότερος σύμμαχος των δραστήριων γεωργών που θέλουν να επενδύσουν. Θέλουν να, να επενδύσουν στο μέλλον τους. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Τώρα θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ορισμένα σημεία στην παρέμβασή μου. Σε έξι. Μία σύντομη εισαγωγή, μία διαπίστωση των καινούριων στοιχείων της νέας κατάστασης, ε, της πρόκλησης της αγροτικής ανάπτυξης. Θα αναφερθώ στις, ε, στη διαδικασία της μεταρρύθμισης ε, που ξεκίνησε από το 1992 και κάθε πενταετία είχαμε σχεδόν νέα μεταρρύθμιση. Και είναι πολύ δύσκολο να γίνονται συνέχεια αλλαγέ, γιατί δεν μπορούν οι επιχειρηματίε να λάβουν αποφάσει για το μέλλον. Και έτσι αποδυναμώνεται ο κλάδο. Και ακριβώ επειδή υπάρχει πολύ χαμηλή κοινωνική υποστήριξη και η κοινωνική εντύπωση των γεωργών αυτή τη στιγμή είναι έθραυστη, ευάλωτη. Και δεν μπορούμε να ζητήσουμε κρατική ενίσχυση για ένα κλάδο που έχει ε, ευάλωτη τέτοια κοινωνική εικόνα. Γιατί οι πολιτικοί θύνοντες είναι ευαίσθητοι ως προς τη γνώμη των ψηφοφόρων και οι περισσότεροι ψηφοφόροι είναι αστεί, ε, μένουν σε αστικά κέντρα που αγοράζουν ε, το γάλα σε τετραμπρίκ στα σούπερ μάρκετ. Και αυτοί έχουν αρνητική γνώμη για του γεωργού. Πώ λοιπόν οι πολιτικοί θύνοντε να υποστηρίξουν αυτού του Γεωργού που δεν χαίρουν τη γενική εκτίμηση του κοινού. Θα μιλήσω λοιπόν για όλα αυτά τα θέματα. Ε, για το γενικό σενάριο της ε, ανταγωνιστικότητας, ε, για τις πρόσφατες κρίσεις, για τις περίκοπες στον προϋπολογισμό και θα καταλήξω κάποια συμπεράσματα. Η σημερινή κατάσταση πάντως είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είχαμε από το 1958. Η Ευρώπη του 2009 είναι τελείως διαφορετική από την Ευρώπη του 1998. Επίσης, Οι κοινωνικές απαιτήσει των τελευταίων χρόνων τι διαφορές είχαν με τις κοινωνικές απαιτήσει της δεκαετίας του 60 ή με τα βουνά βουτύρου και τις λίμνες γάλακτος με τα τεράστια πλεονάσματα σε γεωργικά προϊόντα της Ένωσης. Δεύτερον, πώς ερμηνεύει και πώς αναλύει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις νέες κοινωνικές απαιτήσει και πώς δρομολογεί τις απαντήσεις απέναντι στις ανάγκες αυτές. Τι μπορεί σήμερα να προσφέρει ο γεωργικός κόσμος για να ενισχύσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ας μην ξεχνούμε ότι για το θέμα αυτό, σε μεγάλο βαθμό, η ευρωπαϊκή οικοδόμηση ήταν κοινή γεωργική πολιτική, ήταν γεωργία. Γιατί η γεωργία ήταν η μόνη καλύβα που χτίστηκε με κοινοτικά τούβλα. Ήταν η πεμπτουσία δηλαδή του ευρωπαϊκού οράματος και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Και η Ευρώπη ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τη γεωργία, με την αγροτική ανάπτυξη, με τον τρόπο διατροφής μας. Και φυσικά υπάρχει και ένας κοινωνικός χαρακτήρας στη διατροφή. Διατροφή δεν είναι μόνο οι θερμίδες που καταναλώνουμε. Υπάρχει και μια κοινωνική διάσταση. Δικαιολογείται λοιπόν μια κοινή γεωργική πολιτική στη, στη νέα πραγματικότητα του 2013. Άλλωστε υπάρχει και απειλή για σημαντικές δημοσιονομικές περικοπές και μεγάλη ανταγωνιστικότητα άλλων πολιτικών. Το σημερινό σενάριο είναι πολύ διαφορετικό από το σενάριο του παρελθόντος. Αυτό είναι γνωστό. Οι έξι χώρες ιδρυτές Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο ήταν λίγες, αλλά ήταν και παρόμοιες. Είχαν ταυτόσιμε ανάγκε, γι' αυτό και συμφωνούσαν ω προ του στόχους του. Σήμερα έχουμε 27 χώρε με διαφορετικέ ε, κοινωνικέ και γεωργικέ καταστάσει. γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει συνένεση ω προ κοινού στόχου. Αλλά και οι παραγωγικοί τομεί έχουν τελείω διαφορετικά χαρακτηριστικά. Με τα πολεμικά στην Ευρώπη η γεωργία είχε θεμελιώδη ρόλο. Σήμερα η γεωργική οικονομία έχει ένα χαρακτήρα παροχής υπηρεσιών, με εξαίρεση τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία ίσω άλλαξε και η γεωργική κοινωνία, άλλαξε και η ευρωπαϊκή κοινωνία. Έχουμε ένα γυράσκοντα πληθυσμό με πολλές μειονότητες που έχουν δικαιώματα, που αναγκάζουν τις ε, θεσμικά όργανα να θεσπίσουν αλλαγές. Υπάρχουν αλλαγέ και για το έδαφο και για του παραγωγικού τομεί και για τι άλλε περιβαλλοντικέ χρήσει αλλά και για την αναψυχή. Αλλά υπάρχει και το θέμα τη ε, αστικής πίεσης που επηρεάζει τη χρήση της γης. κάποια στιγμή θέλουμε ένα τμήμα των γεωργικών δαπανών να τις αφιερώσουμε στην περιφερειακή πολιτική. Αυτό βέβαια θα ισοστάθμιζε τους προϋπολογισμούς και μερικές χώρες ε, εξυπηρετούνται με κάτι τέτοιο και βολεύονται και συμφωνώ με την κυρία Μπέλα ότι θα ήταν το τελευταίο που θα έπρεπε να εξετάσουμε για να μην πούμε τίποτα άλλο, για τους στόχους. Θα ήταν πάντως πολύ επικίνδυνο κατά τη γνώμη μου και, και κατά τη γνώμη της ομάδας των επιστημόνων που εκπώνησαν την έκθεση να, να βγάλουν τα στοιχεία της περιφερειακής πολιτικής από το κοινωνικό ταμείο της γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης και ανάπτυξη πέθρου. Γιατί πώς θα καταλάβει τις δυσκολίες ο Γεωργός μιας απομονωμένης ζώνης μειονεκτικής που αντιμετωπίζει προβλήματα με την καλλιέργειά του σε μια πολύ αεροκατοικημένη περιοχή 25 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ενώ σε άλλες περιπτώσεις ε, έχουμε στις πόλεις πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού και τελείως διαφορετικές ανάγκες. Αλλάζουν και τα περιβαλλοντικά στοιχεία, αλλάζουν και τα μοντέλα κατανάλωσης και απειλέ συρρήκνωση του προπολογισμού. Εκτό από αυτέ τι εσωτερικέ αλλαγέ, υπάρχουν και εξωτερικέ αλλαγέ. Αναφέρθηκαν οι αλλαγέ από τη Συμφωνία Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου, αλλά και οι δημογραφικές αλλαγές παγκοσμίω. Όλα αυτά έχουν υπέρ και κατά. Σε παγκόσμια κλίματα, κλίμακα έχουμε και τι κλιματικές αλλαγές και το πρόβλημα της ε, ενέργειας, αλλά και την χρηματοπιστωτική και επισητιστική κρίση. Ένα νέο σενάριο προϋποθέτει νέες ανάγκες. Αυτές οι νέες ανάγκες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να καθοριστούν οι νέοι στόχοι. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σε αυτό το νέο σενάριο η Ευρωπαϊκή Ένωση ερμηνεύει και δρομολογεί τις ε, απαιτήσει. Από το 2005 είχαμε τη στρατηγική της Λισαβόνας ε, που ξεκίνησε το 2000 και το 2001-2006 είχαμε τη στρατηγική του Γκέτεμπουργκ που οδήγησαν σε διαφορετικές θέσεις. Μεταξύ των θεσμικών θέσεων η πιο σημαντική ήταν το έγγραφο 2020 που ε, συμπληρώνεται με τέσσερα έγγραφα. Το ένα ετοιμάζεται για δημοσίευση και τα άλλα ήδη κυκλοφορούν από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και τα έγγραφα αυτά ε, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην περιφερειακή πολιτική γιατί μιλούν για τέσσερις σημαντικές προκλήσεις, τη δημογραφική, την περιβαλλοντική, την, και την παγκοσμιοποίηση αλλά και τη χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτές οι τέσσερις προκλήσεις φέρνουν τη Γενική Διεύθυνση ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, σε θέση χάραξης κάποιων πολιτικών. Υπάρχουν και άλλες ε, ανταγωνιστικές πολιτικές. Έχουμε την πολιτική κοινωνικών υποθέσεων και απασχόλησης, περιβάλλοντος, ενέργειας, μεταφορών και κατανάλωσης. Και σε αυτόν τον κόσμο των καρχαριών, όπως είπε και η κυρία Επίτροπος, ε, ποια είναι η θέση της ΚΑΠ. Για πρώτη φορά, και αυτό είναι καινούριο, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός νέων κοινοτικών πολιτικών βρίσκονται σε ανταγωνισμό μεταξύ τους. Και δεν ζητούμε μόνο από την ΚΑΠ να περιορίσει τον προπολογισμό τη, αλλά να ανταγωνιστεί άλλε πολιτικέ που είναι και πιο δραστήριες. Στην Ήπεθρο, όμως, έχουμε μια μεγάλη δύναμη, γιατί καμία άλλη πολιτική, κανένας άλλος δικαιούχος πολιτικής, δεν είναι ικανός να συγκεντρώνει όλες τις νέες προτεραιότητες και όλες τις νέες προκλήσεις Ευρώπης ταυτόχρονα. Αυτό το κάνει η υπέθρο, συγκεντρώνει όλες αυτές τις προκλήσεις. Άλλωστε το 90% της Υπέθρου ε, έχει εγκάρσια χαρακτηριστικά για όλες τις πολιτικές. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, για να αναγνωριστεί η σπουδαιότητα της Υπέθρου. Για μια πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και πολιτική υπαίθρου, γιατί θα πρέπει από κοινού να τα συνδυάζουμε αυτά, να μην εξετάζουμε την γεωργία άσχετα με την αγροτική ανάπτυξη ή την ύπεθρο. Είναι αλληλένδετα τα δύο θέματα. Η χρηματοδότηση μερικές φορές βέβαια είναι διαφορετική για παρόμοια θέματα και ίδια για άσχετα θέματα. Αυτό φαίνεται ότι και στο διαγνωστικό έλεγχο. Θα πρέπει όμως να λαμβάνουμε υπόψη από κοινού τη γεωργική ανάπτυξη με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει συνένεση για την συνέχιση της ΚΑΠ. Πολλοί μιλούν για σημαντικές ερυκνώσεις και περικοπές του προϋπολογισμού του, της ΚΑΠ, αλλά συνένεση δεν υπάρχει, φημολογίες μόνο. Και φυσικά στην περίοδο των ισχνών αγελάδων όλοι γίνονται τσιγκούνιδες. Και ούτε καν η δέσμευση σταθερότητα τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση δεν τηρείται. Οπότε καμία χώρα ε, δεν θέλει να ακούσει για περισσότερα κονδύλια στη Γεωργία. Πάντω, ο μόνο τρόπο για να νομιμοποιηθεί μια κοινή πολιτική αγροτική ανάπτυξη είναι να είναι αποτελεσματική αυτή η πολιτική για τα επόμενα χρόνια. Οπότε θα πρέπει να αποδείξει την προστιθέμενη αξία της και μάλιστα την προστιθέμενη ευρωπαϊκή της αξία. Αυτό είναι εύκολο να το λέμε, αλλά δύσκολο να το εφαρμόζουμε. Μία μεταρρύθμιση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης ξεκίνησε ήδη με τη μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ και φτάνει μέχρι το διαγνωστικό έλεγχο. Και βλέπουμε μία σύγχυση και με τα μία, τα διαρθρωτικά, το πρώτο που έγινε δύο, το ΦΕΟΓΑ, μετά το ΦΕΟΓΑ εγγύησης. Είχαμε το ΦΕΟΓΑ προσανατολισμός και μετά το ΦΕΟΓΑ εγγύησης. Το 1992 με τις πρώτες ε, κοινωνικο-οικονομικές ε, οδηγίες ε, δεν ήταν καν διαρθρωτικό ταμείο το ΦΕΟΓΑ, αλλά μετά με τις μεταρρυθμίσεις το 89 προέκυψε το ΦΕΟΓΑ προσανατολισμός διαρθρωτικό, αλλά όχι το ΦΕΟΓΑ εγγύησης. Και στο πρόγραμμα του 2000, ακόμη και το ΦΕΟΓΑ εγγυήσει, έγινε διαρθρωτικό ταμείο για τις ζώνες όχι του στόχου 1 και άρχισε να χρηματοδοτεί πράγματα που δεν ήταν μόνο ρύθμιση αγορά ή στήριξη του εισοδήματο. Είναι πολύ συγκεχημένα όλα αυτά τα πράγματα. Ακόμη και για τον επαγγελματία, ακόμη και για τον ειδήμονα, το τοπίο είναι θολό. Και φαντάζομαι για έναν απλό φορολογούμενο όλα αυτά ακούγονται αποκρυφιστικά. ε, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Ε, ε από τη μια μας δηλητηριάζουν, από την ε, άλλη είναι ασαφή αυτά που προτείνουν. Θέλουμε όμως μια πρόταση που να είναι σαφής και εύληπτη για τον απλό πολίτη. Και όχι μόνο να είναι εύληπτη, αλλά και ενδιαφέρουσα για τον πολίτη, για να καταλάβει ο πολίτης ότι αυτή η, η πρόταση σχετίζεται και με το μέλλον του. Ό,τι αφορά την αποσύνδεση, Υπάρχει μια πρώτη περίοδος μέχρι τη μεταρρύθμιση του 1992 που δεν υπάρχει ανάγκη για αποσύνδεση. Γιατί δεν είχε περιληφθεί τότε το γεωργικό κατά κεφάλαιο στις διαπραγματεύσεις της τότε ΓΚΑΤ. Από το 1992 μέχρι το 2003 όμως εφαρμόζεται μία αποσύνδεση από την παραγωγή. Και εκεί έχουμε ένα τμήμα της ιστορικής ευθύνης. Και μετά την ενδιάμεση αναθεώρηση του 2003 έχουμε αποσύνδεση και από το προϊόν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα έχουμε κάποια κονδύλια που είναι αποσυνδεδεμένα από το παρελθόν. Αυτό μου θυμίζει κάποιους ελιγμούς που γίνονται στο τσίρκο όταν κάποιος είναι σχηνοβάτης ή κάποιοι που κάνουν περίεργες, ε, ε, ε περίεργες ασκήσεις ε, στα τραπέζια χρειάζεται να κάνουν διάφορες κουλουτούμπες. Και μάλιστα βρίσκονται μονίμως στον αέρα. Αυτό μου θυμίζει κάπου. Σαν να χάθηκε η επαφή με τον οφάλιο λόρο. Δεν έχει εξασφαλιστεί συνέχεια με το νέο σενάριο. Ενώ ταυτόχρονα ε, χάσκουν οι καρχαρίες των άλλων ανταγωνιστικών πολιτικών. Όλη αυτή η σύγχυση λοιπόν, όλο αυτό το κομφούζιο, τι είναι, είναι η αγροτική ανάπτυξη, είναι η πολιτική της υπαίθρου. Όταν κάποιος ακούει τη όρο ανάπτυξη, θεωρεί ότι χρησιμεύει για ανάπτυξη, ότι είναι κάτι που εξελίσσεται. δεν μπορεί να καταλάβει ο πολιτή ο απλός πολίτης κάποια μέτρα τη ΚΑΠ. Και όταν ακούει ανάπτυξη θέλει πραγματικά ανάπτυξη υπαίθρου και τα μέτρα που προορίζονται για την ανάπτυξη υπαίθρου να την αναπτύσσουν και να μην περιλαμβάνονται στην ανάπτυξη υπαίθρου μέτρα που είναι άσχετα με την ανάπτυξη υπαίθρου. Ε, λοιπόν, με είπα για τον καθηγητή ε, Μπάκουελ που ήταν ε, καθηγητής του του CLA, τον ξέρω από παλιά. Μίλησε λοιπόν για όλα αυτά τα θέματα μεταξύ της διαφοράς λειτουργίας του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα. Τα τελευταία χρόνια όμως όλα αυτά τα όρια των δύο πυλώνων έχουν γίνει πολύ ρευστά και συγκεχημένα. Το σημερινό μας όμως θέμα είναι η γεωργική πολιτική μετά το 2013. Και ο κύριος Σαντελέ και ο κύριος Πάκολ αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για χρήματα αν δεν συμφωνήσουμε προηγουμένω για του στόχου. Γιατί πρώτα θα καθορίσουμε του στόχου και μετά θα προβλέψουμε του πόρου για να του χρηματοδοτήσουμε. Επίση, θα πρέπει να γίνει μια ανακατανομή των δαπανών μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα, αλλά και μεταξύ χωρών. Γιατί αυτό, ε, γι' αυτό παραπονιούνται οι πολίτε, ότι δεν είναι οι πλέον άποροι αυτοί που λαμβάνουν τα περισσότερα κονδύλια, ούτε αυτοί που τα χρειάζονται περισσότερο. Α μην ξεχνούμε ότι ορισμένες από τις αποφάσεις που θα λάβουμε ίσως έχουν ανεπανόρθωτα αποτελέσματα. Και αυτά τα επανόρθωτα αποτελέσματα, ιδιαίτερα στη γεωργία που στηρίζεται με τους φυσικούς κύκλους, που είναι πιο ε, μακροπρόθεσμοι από τους βιομηχανικούς, είναι δύσκολο να λαμβάνουμε τέτοιες αποφάσεις ανεπανόρθωτες, γιατί δεν μπορούμε να ανακτήσουμε μερικέ φορέ τα αποθέματα. Θα χρειαστούν ολόκληρε γενιέ και προσπάθειε γενεών για να διορθωθεί μια τέτοια απόφαση. Ορισμένε άλλωστε αποφάσει και ορισμένα πράγματα γίνονται καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ό,τι σε εθνικό. Επίση, έχουμε την πολυλειτουργικότητα, τα δημόσια αγαθά, τα επιχειρήματα που νομιμοποιούν το δεύτερο πυλώνα. Οι αλλαγέ ε, είναι πολύ σημαντικέ. Γι' αυτό θα πρότεινα ε, μία μεταρρύθμιση σε δύο φάσει. Στην πρώτη φάση μεταβατικά μέτρα, πολύ πιο έφεπτα για τα κράτη-μέλη, που θα έχουν όμως ήδη τη φιλοσοφία των συμβάσεων και σε δεύτερη φάση πιο προηγμένη και μεσοπρόθεσμη. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπε η Επίτροπος Φίσερ Μπέρλ το 2005 μετά από μια συμφωνία του Συμβουλίου Γεωργίας σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Γεωργίας του 1997. Νομίζω ότι ήταν πολύ εύστοχη αυτή η φράση της Επιτρόπου Φίσερ Μπέλ που μίλησε για τα διάφορα είδη γεωργίας και τους διάφορους ρόλους που απαιτεί από τη γεωργία η ευρωπαϊκή κοινωνία. Αυτό αναφέρθηκε πρώτα το 1997 και μετά το 2005. Έφυγε όμω η επίτροπο και δεν πρόλαβα να τη ρωτήσω αν τώρα με το νέο σενάριο και με την κρίση θα επέμεινε σε αυτή τη θέση που σχετίζεται και με το επίπεδο ευημερία που απαιτούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Για να ετοιμάσω το πόνημά μου διάβασα πολλή βιβλιογραφία και για τα σενάρια του 2020 πολλών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων και διάβασα πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες από την Ρουλάλης, <laughs> πιστεύω ότι υπάρχουν δύο άξονες για την ανάλυση της νέας πολιτικής. Έχουμε ένα επίπεδο ρύθμισης ε, οριζόντια και κόρυφα ένα επίπεδο απελευθέρωσης. Και όλα αυτά γίνονται είτε σε διμερές επίπεδο είτε σε πολυμερές επίπεδο. Και υπάρχει το θέμα της περιφερειοποίησης. Και μάλιστα σε με μια πιο εδαφική προσέγγιση θα αντιλαμβανόμασταν καλύτερα την αγροτική ανάπτυξη. Σε αυτή την πρώτη μεταβατική φάση θα θέλαμε ένα σπίτι παρόμοιο αυτό του Φεντέρ, αλλά παρόμοια αλλά διαφορετική στην ουσία της. Έχουμε τρεις άξονες, τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο, που έχουν τα ίδια, τις ίδιες ονομασίες, αλλά ο τρόπος διαχείρισης των αξώνων είναι διαφορετική. Επίσης ε, υπάρχει ένα υπόθεμα μόνος προς τις συμβάσεις των περιφερειακών σχεδίων και ένας προϋπολογισμός προς το συλλογικό ώστε να υπάρχει συλλογική ευθύνη απέναντι στους φυσικούς πόρους και να αναλαμβάνουν ε, αυτή τη συλλογική ευθύνη οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Και υπάρχει και ο στρατηγικός στόχος. Ό,τι αφορά τις ελάχιστε, τα ελάχιστα ποσοστά προτιμώ να αυξηθούν για τον πρώτο άξονα 10 με 15%, για το δεύτερο άξονα μέχρι 30% και για το τρίτο άξονα μέχρι 15%. Και υπάρχει και ένας ηγετικό άξονας που δεν συνοδεύεται από ποσόστοση. Γιατί τη γνώμη μου είναι εγκάρσιος αυτός ο ηγετικό άξονας, όχι οριζόντιος. Δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά στις οθόνες. Αυτός ο άξονας leader είναι η μεθοδολογία του Λίντερ και ο άξονας 1 και 2 εξασφαλίζουν τουλάχιστον 5% των δύο αξώνων γίνεται με συμμετοχική μεθοδολογία. Αλλά σε πιο προηγμένη φάση εγώ θα ανέβαζα τα ποσοστά απέτηση συλλογική δράσης στους δύο πρώτους άξονες. Σε ό,τι αφορά το μέσο και μακροπρόθεσμο θα προτιμούσα κοινό κορβανά. Στον πρώτο ε, πυλώνα μηχανισμούς ρύθμισης των αγορών και στο δεύτερο πυλώνα νέο χρηματοπιστωτικό μηχανισμό, ένα ευρωπαϊκό ταμείο γεωργικής ε, ανάπτυξης και ανάπτυξη πέθρου ή όπως άλλως θέλετε πείτε το και ένα άθροισμα των δύο. Επίσης θα πρέπει να αφαιρεθούν οι δημοσιονομικές περικοπές που σίγουρα θα γίνουν, αλλά υπάρχει δυνατότητα κρατικής συγχρηματοδότηση. Άλλωστε, οι πιο εύρεστες οικονομίες ε, έχουν αντιληφθεί την ανάγκη της συγχρηματοδότησης. Το θέμα είναι σε τι βαθμό, με τι ποσοστό θα γίνεται η συγχρηματοδότηση, προκειμένου να μην ε, απολυστεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και τα κονδύλια αυτά θα διαλυθούν σε δύο τμήματα, σε ένα εγκάρσιο οριζόντιο και σε ένα περιφερειακό. Στο περιφερειακό πρόγραμμα ε, θα υλοποιούνται στόχοι αναπτυξιακοί. Και όπω λέει και η αναπτυξιακή θεωρία της οικονομίας, συγκεντρώνει κάποιες δραστηριότητες ε, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικότητα, ανάπτυξη και βιωσιμότητα. Το οριζόντιο πρόγραμμα ασχολείται με πιο γενικά προβλήματα. Έτσι, τα κονδύλια αυτού του ταμείου θα χρηματοδοτούν πρώτα ένα οριζόντιο πρόγραμμα για τη διαχείριση των κινδύνων, της επισητιστικής ασφάλειας αλλά και των χρηματοπιστωτικών κινδύνων ή των κινδύνων που απορρέουν από την παγκοσμιοποίηση. Αυτό το πρόγραμμα θα έχει οριζόντιο χαρακτήρα και θα οδηγούσε στην ε, θέσπιση κάποιων δικτύων ασφαλείας και στα, στα προγράμματα τα περιφερειακά θα είχαμε κατά αποκοπή ποσά flat rate για όλες τις μελλοντικέ δραστηριότητες προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το κόστος της νέας γεωργίας. Και έχουμε και τη χρηματοδότηση για την εξασφάλιση μιας ευημερία. Μας ενδιαφέρει φυσικά όχι μόνο η ανταγωνιστικότητα αλλά και το περιβάλλον. Αυτό είναι παρόμοιο προς, τους στόχους. Την αποτελεσματικότητα, την ισότητα, την ισοτιμία και τη βιωσιμότητα. Αυτό ισχύει και για την Ήπεθρο και για τη Γεωργία. Γιατί όταν λέμε ισοτιμία εννοούμε ισότητα και δικαιοσύνη. Αυτά ανήκουν στο δεύτερο πυλώνα. Και ό,τι είναι αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα ισχύει για τις μη αγροτικές δραστηριότητες και τις αρμοδιο... δραστηριότητες βιοπικιλότητας. Στην έκθεση του 2008 για τη γεωργική ανάπτυξη είχαμε πολύ ενδιαφέροντες χάρτες για τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν σε θέματα διαφοροποίησης και παραγωγικότητας. Στις περιοχές με μεγαλύτερο κοινωνικό κεφάλαιο και μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη υπάρχει και μεγαλύτερη δυνατότητα διαφοροποίησης. Ενώ στις περιοχές που έχουμε πιο τη γεωργία και υπάρχουν παντού στην Ευρώπη και στις παλιές και στις νέες χώρες και στο βορρά και στο νότο, εκεί η διαφοροποίηση και η παραγωγικότητα δεν πρόκειται να δημιουργήσουν επιπλέον εισόδημα. Και φυσικά αν λειτουργήσουν αυτά χρόνο με το χρόνο θα δούμε πώς ε, οι συμβάσεις θα αντιμετωπίσουν, θα αντικαταστήσουν το καταποκοπήν ποσό. Και για να φτάσουμε στα συμπεράσματα. Δύο ιδέες ως προς την πρώτη ερώτηση. Τι μπορεί να προσφέρει, τι να προσφέρει σήμερα η Ήπεθρος για να ενισχυθεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Μία κοινή απάντηση σε όλες τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να συμβάλλει φυσικά στην ε, συνοχή και στην ισορροπία μεταξύ των διαφόρων ε, αγροτικών περιοχών. Ε, δικαιολογείται μια κοινή γεωργική πολιτική για την εποχή μετά το 2013. Νομίζω ότι οι υπεθρός, οι αγροτικές ζώνες μπορούν να δεσμευθούν και να γίνουν μια πραγματική ατμομηχανή, ένας κινητήριος μοχλός της διαδικασίας ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Γιατί η Ευρώπη στην αρχή είχε γεωργικό χαρακτήρα και εξυπηρετούσε κυρίως διατροφικές ανάγκες. Με τις νέες όμως προκλήσεις, μια ενωμένη ισχυρή και μεγάλη Ευρώπη θα μπορούσε να αναλάβει τις νέες προκλήσεις με τη συνεργασία των αγροτικών ζωνών. Τώρα, είναι όλα αυτά ένα όνειρο? Η Ήπεθρος μπορεί να απολαύσει μια πολιτική αγροτικής ανανάπτυξης που θα έχει την υποστήριξη και της ευρωπαϊκής κοινωνίας στο μέλλον. Αυτό δεν είναι όνειρο μπορεί να γίνει και πραγματικότητα. Ελπίζω να σα έπεισε και να σα τα πέδειξα με αυτά που είπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο, τον Ράμος. Θα περάσουμε στην ε, επόμενη παρέμβαση πάρα γιατί καθυστερήσαμε λίγα εκεί προηγουμένω και αν θέλουμε να έχουμε και λίγο χρόνο για τη συζήτηση, καλύτερα θα τον ακούσουμε τώρα την επόμενη παρέμβαση. Ο κύριος Βαλάντα Ζάντε θα μας παρουσιάσει τις δημοσιονομικές πτυχές των πληρωμών της νέας ε, κοινής αγροτικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την ε, μετά το 2013 κατάσταση. Κύριε Ζαντ, εάν θέλετε, σας ακούμε. Να, να πάρετε το λόγο Members of the Parliament, ladies and gentlemen. Αγαπητοί βουλευτές, κυρίες και κύριοι, ε, νομίζω ότι καταρχάς θα έπρεπε να μιλήσουμε πρώτα για τους στόχους και μετά για τα δημοσιονομικά. Ε, το κακό βέβαια όταν μιλάς τελευταίος είναι ότι το κοινό σου έχει κουραστεί λιγάκι. Ε, θα ήθελα όμως να δω τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική γωνία και ελπίζω να με ακούσετε. Το πρόβλημα με τα δημιουργικά σενάρια για τον προπολογισμό τη ΚΑΠ είναι ότι έχουμε πολλού σημαντικού εταίρου, παράγοντε, του οποίου ε, δεν γνωρίζουμε καλά, δεν μπορούμε να του προσμετρήσουμε και δεν μπορούμε να δούμε πώ θα αλληλεπιδράσουν. Ε, Προ το παρόν, λοιπόν, ε, μπορούμε μόνο να μιλήσουμε με σενάρια. Ε, να πούμε ότι έτσι πιστεύω ότι θα ξοδευτούν τα χρήματα, αλλά αυτό εξαρτάται και από τι πολιτικέ προτάσει. Βλέπετε τα θέματα σε, αυτό σε αυτή τη διαφάνεια που θα θίξω. Καταρχάς, το πρώτο θέμα είναι η χρηματοδότηση και η ύπαρξη κονδυλίων. Θα ήθελα να ε, κάνω μια αναθεώρηση της πρόσφατης ε, οικονομικής κρίσης που θα έχει ε, σοβαρότερε επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΚΑΠ. Θα πιέσει τους εθνικούς προϋπολογισμούς και θα τροποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε δημόσιες δαπάνες. Με βάση την Κομισιόν, τα ελλείμματα των προϋπολογισμών θα αυξηθούν ε, σε 6% το 2009 και 7,3% το 2010. Και 20 κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή ε, διώκονται για παραβίαση του Συμφώνου Σταθερότητας. Ε, με αυτόν τον τρόπο το 2008 θα έχουμε το λόγο ε, ελλείμματος, χρέους μάλλον, προς ΑΕΠ, 60% ε, το 2008, 70% το 2009, 80% ε, το 2010. Αν η ανάπτυξη επανέλθει στα επίπεδα πριν την κρίση και διατηρήσουμε τις σημερινές πολιτικές, τότε το χρέος θα φτάσει το ΑΕΠ το 2013 και εν συνεχεία τα επόμενα χρόνια θα το ξεπεράσει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι απίθανο ότι τα κράτη-μέλη ε, τα οποία ιστορικά ήταν απρόθυμα να δώσουν περισσότερα κονδύλια θα γίνουν πιο γενναιόδωρα. Μπορούμε να ελπίσουμε ότι ε, ίσως με τους, νέους, με τους ίδιους πόρους ή με το σύστημα εμπορίας ε, των εκπομπών ε, θα έχουμε νέες δυνατότητες. Αλλά όλα αυτά είναι μακροπρόθεσμα προγράμματα και δύσκολα θα επηρεάσουν τις επόμενες οικονομικές προοπτικές, χρηματοδοτικές προοπτικές. Έπειτα το θέμα είναι τι μερίδιο του προϋπολογισμού θα πάει στην ΚΑΠ. Ε, προφανώς υπάρχουν και άλλες ανάγκες και συχνά υπάρχει, υπάρχουν διεκδικήσεις ε, για το κλίμα, για την ενέργεια κτλ ενώ μπορεί να υπάρξει ουσιαστική μείωση για την ΚΑΠΑ ε, από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Μπορεί αυτοί που υποστηρίζουν ένα ευρύ προϋπολογισμό να χάσουν. Τα κράτη-μέλη, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν ουσιαστικά αυτή την αύξηση, ε, μπορεί να ε, μην θεωρήσουν πλέον ότι υπάρχουν λόγοι για τέτοια αύξηση του προϋπολογισμού. Αυτά τα κράτη-μέλη τα οποία εποφελούνται από τη σημερινή κλίδα κατανομής μπορεί να χάσουν, ενώ πολλά κράτη-μέλη θα δουν ότι θα έχουν μεγαλύτερο μερίδιο ε, του προϋπολογισμού, παρόλα αυτά θα ζητήσουν μείωση του προϋπολογισμού την ΚΑΠ. Ε, παραδείγματος χάρη Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλα κράτη-μέλη ε, προτιμούν να πάρουν ε, περισσότερα κονδύλια από τα διορθωτικά ταμεία, παραδείγματος χάρη οι, Ανατολ... οι χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Όλα αυτά τα θέματα είναι περίπλοκα και Δεν μπορούμε να παραμένουμε σε γενικόλογες ε, διακηρύξεις. Όταν σκεφτόμαστε τις μελλοντικέ ανάγκες ε, χρηματοδότησης, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τους στόχους της πολιτικής. Ας εξετάσουμε ε, τα, τους τρεις στόχους της ΚΑΠ και ας δούμε πόσα λεφτά πρέπει να επενδύσουμε σε ό,τι αφορά την τη στήριξη του εισοδήματος. Υπάρχουν ε, διάφορες επικρίσεις ε, ότι οι κοινωνικές πολιτικές θα πρέπει να συνδέονται ε, με, τα, με την ευρωστία των οικοκυριών και όχι με άλλα κριτήρια, αν υπάρχει ας πούμε ιδιοκτησία της γης. ορισμένοι ας πούμε γεωργοί ούτως ή άλλως έχουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία ή είναι πλούσιοι. οι φτωχοί γεωργοί συχνά εποφελούνται λίγο από τις ενιαίες πληρωμές και οι κοινωνικέ ε, πολιτικέ δεν θα πρέπει να πληρωθούν, λένε κάποιοι άλλοι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τέλεια χρηματοδότηση λοιπόν σε αυτήν την περίπτωση είναι μηδενική. Σε ό,τι αφορά την επιστηστική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μάλλον απίθανο να υπάρξουν τέτοιε ελλείψει ε, τροφή. Καταρχά, η παραγωγή μα είναι αρκετά μεγάλη και επίση ε, με πιο εντατικέ μεθόδου καλλιέργεια μπορούμε να καλύψουμε τι μεγαλύτερε ανάγκε αν πετάμε λιγότερα φαγητά, ε, θα έχουμε περισσότερα στο πιάτο μας, σε περίπτωση που έχουμε λήψει. Επίσης, έχουμε αρκετή, αρκετά μεγάλη αγοραστική δύναμη, α, ακόμη, για να καλύψουμε τι ανάγκε μα, ακόμη και όταν είναι ψηλά οι παγκόσμιες τιμές. Ε, δεν χρειάζεται να δώσουμε πολλά κονδύλια στην επιστημιστική ασφάλεια. Ε, θα πρέπει να διατηρήσουμε το νερό, βιοπικιλότητα και τη γενετική ποικιλία των φυτών σε ό,τι αφορά τα δημόσια αγαθά. Ε, τα συμπεράσματα για τον προϋπολογισμό λένε ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να γίνεται εκεί όπου υπάρχει προσθέμενη αξία και ο κοινοτικό προπολογισμό θα πρέπει να εξασφαλίσει την παροχή των δημοσίων αγαθών. Όμω, το ποσό τη χρηματοδότηση που χρειάζεται για την προώθηση των ε, δημοσίων αγαθών είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Ε, καθορίζεται προφανώ από, το τι είναι, από, τον, από τον ορισμό του δημοσίου αγαθού. Μπορούμε να πούμε ότι παραδείγματο χάρη ε, είναι καλό να έχουμε να διατηρήσουμε το παραδοσιακό ας πούμε, τοπίο, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα προσελκύσουμε τουρίστες. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι πρόθυμη να κάνει κάποιες συλλογικέ επενδύσεις. αυτή την Τρίτη θα δημοσιευθεί μία μελέτη ε, για αυτά τα θέματα. Όταν εντοπίσουμε τους ε, στόχους, εν συνεχεία, τους στόχους και τι είναι τα δημόσια αγαθά, θα πρέπει να δούμε πώς θα τα εξασφαλίσουμε. Επίσης, Κάτι άλλο που θα πρέπει να δούμε είναι αν θα αντιμετωπίσουμε τη γεωργική και δασοκομική γη με πιο δίκαιο τρόπο. Αν η ΚΑΠΑ χρηματοδοτήσει περισσότερα, χρειάζεται περισσότερα δημόσια αγαθά, τότε χρειάζεται και μεγαλύτερη χρηματοδότηση. όσο ρυθμίσουμε πιο αποτελεσματικά τους στόχους και βρούμε άλλους πόρους, τόσο λιγότερες ε, επιδοτήσεις θα χρειαστούμε για τη γεωργία. Πάντως, ε, το επίπεδο χρηματοδότησης ε, των δημοσίων αγαθών δεν είναι γνωστό ακόμα. Εξαρτάται από την ποιότητα και ποσότητά τους. Και επίσης, πρέπει να δούμε τι θα πληρώσουν και οι κυβερνήσεις για να πετύχουν αυτά τα δημόσια αγαθά, εάν επιθυμούν να τα αποκτήσουν. Το, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι εύκολη, γιατί πάρα πολλά στοιχεία το προσδιορίζουν, παραδείγματο χάρη α, τιμές, τις αγορές τιμές, ε, δασμολογικές Ε, ε, δασμολογικά έσοδα, ε, διοικητικό κόστος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κτλ. Πέρα τώρα από τον προσδιαρισμό των στόχων θα πρέπει να δούμε το θέμα της χρηματοδότησης μελλοντικής ΚΑΠ. Παρά την, το μακρό παρελθόν της, η βασική αρχή της αλληλεγγύης, δηλαδή 100% χρηματοδότηση από το κοινοτικό προπολογισμό, είναι δύσκολο να διατηρηθεί. Ε, ένα επιχείρημα είναι ότι η χρηματοδότηση της ΚΑΠ ε, βοήθησε και ευνόησε συγκεκριμένα κράτη-μέλη και περιοχές. Η ΚΑΠ, λένε κάποιοι, θα πρέπει να εξασφαλίζει ε, και να βοηθάει την αναδιανομή του πλούτου. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν την ΚΑΠ σε συνδυασμό και με τους στόχους των διαρθρωτικών ταμείων. Υπάρχουν αρκετά προνεκτήματα στη συγχρηματοδότηση. Καταρχάς, ε, δίνονται κίνητρα στα κράτη-μέλη για να χρησιμοποιήσουν ε, με λογικό τρόπο τα κοινοτικά κονδύλια. Τα κράτη-μέλη θα διαχειριστούν τα κονδύλια πιο αποτελεσματικά και θα έχουν μεγαλύτερη ωφέλη για, εμένο, για την υλοποίηση ενός στόχου αν συμμετέχουν στο κόστος. Η συγχρηματοδότηση ε, δίνει στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να επηρεάσει περισσότερα τα πράγματα και να διαμορφώσει πολιτικές με βάση τις δικές της προτεραιότητες. Ε, επομένως, μπορούμε, θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε τη συγχρηματοδότηση σε όλη την ΚΑΠ. Αλλά όμως τα κράτη-μέλη είναι διαιρεμένα εδώ. Και τα συμπεράσματα του, της του προϋπολογισμού λένε ότι θα πρέπει να έχουν περισσότερα, περισσότερη ευθύνη τα κράτη-μέλη και οι άμεσες ε, ενισχύσεις θα πρέπει να συγχρηματοδοτούνται. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε τόσο ώστε να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση των ε, αποφάσεων και των πολιτικών. Θα πρέπει να προωθήσουμε τα δημόσια αγαθά τα οποία έχουν διασυνοριακή διάσταση παρά εκείνα τα οποία παραμένουν στο εσωτερικό μία και μόνη χώρα. Η διάκριση μεταξύ τριών ειδών προγραμμάτων στο δεύτερο πυλώνα δεν είναι επιτυχή και ο βαθμό ε, συγχρηματοδότηση δεν είναι ο επιθυμητό. Δεν είναι αρκετά υψηλό. Τώρα, ε, διασύνδεση με άλλες πολιτικές αυτό θα έχει πολύ σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις. Με βάση τη σημερινή διάρθρωση, ε, η διασύνδεση της πολιτικής συνοχής και ανάπτυξη πένθρου ε, βοηθάει την πιο εύλογη εφαρμογή. Ε, όταν η πολιτική έχει σαν σκοπό την βιώσιμη χρήση της γης, αυτό βοηθάει και επίσης ο όρος γεωργική πολιτική είναι παραπλανητικός. Δίνει την ε, εντύπωση ε, στους ε, γεωργούς ότι τα δικά τους λεφτά χρησιμοποιούνται για τη δασοκομεία, για το περιβάλλον, για άλλους σκοπούς. Καλό θα ήταν όλες οι πολιτικές να ομαδοποιηθούν, πολιτικές που αφορούν την βιώσιμη χρήση της γης και να μετονομάσουμε τις πολιτικές αυτές. Με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξουν και οι προσδοκίες για τους στόχους ε, των πολιτικών. Ε, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Κομισιόν θέλει να αλλάξει άρτενο ο κοινωτικός ε, προϋπολογισμός. Ε, επομένως, διάφοροι, διάφορα κεφάλαια των δημοσιονομικών προοπτικών θα περιοριστούν και θα υπάρξει ε, μεγαλύτερος κατακαιρματισμός σε διάφορες πολιτικές, ούτως ώστε να καλυφθούν καλύτερα οι ανάγκες. Ακόμη και αν σας αρέσουν αυτά τα σχέδια συμπερασμάτων και πολλοί φαίνεται ότι δεν ε, συμφωνούν, νομίζω ότι αντανακλούν τις ε, βασικές απόψεις μεταξύ πολλών και ακόμα και πολλών επιχειρηματιών και νομίζω θα πρέπει να τις, λάβουμε, να τις πάρουμε σοβαρά υπόψη. Οι στρατηγικές μετάβασεις Ούτως ή άλλως θα χρειαστούμε στρατηγικές μετάβασεις ε, προς μια μικρότερη ΚΑΠ ε, που είναι πιο καλά προσαρμοσμένη προς τα δημόσια αγαθά. Θα μπορούσαμε, παράδειγμα, χάρη, να έχουμε μια γραμμική μείωση της ενιαίας πληρωμής. Είναι πολύ πιο αποτελεσματική κοινωνικός πώς ε, και θα είναι λιγότερο δαπανηρή. Αυτή η μικρότερη ενιαία πληρωμή θα μπορούσε να βασιστεί στα δικαιώματα που έχει ο καθένας. Βέβαια, με μια γραμμική μείωση. Θα πληρώνουμε λιγότερο στους απλούσιους ε, και θα πληρώνουμε περισσότερα σε αυτούς που εξαρ... στα νοικοκυριά που εξαρτώνται από τη γεωργία. Πέρα από κάποιο ε, κατόφλι, δεν θα δίνεται καμία πληρωμή. Ένα άλλο μέτρο που θα μπορούσε να μειώσει το βάρος ε, σε αυτή τη μεταβατική φάση της ΚΑΠ θα ήταν να ε, συμπληρώσουν ε, τα ποσά οι κυβερνήσεις. Μια και τα συστήματα ούτως ή άλλως είναι μία, μία ακριβή, ε, δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Νομίζω ότι το βασικό είναι να μην ξεχνάμε ποιος είναι ο μελλοντικός στόχος της ΚΑΠ αυτό θα μας επιτρέψει να είμαστε τολμηροί σε σχέση με τους στόχους και πιο ευέλικτοι σε σχέση με τις, τις μεταβατικές αυτές πληρωμές. Είμαστε αβέβαιοι πάντως για την διαθεσιμότητα των ε, κονδυλίων. Νομίζω είναι πολύ να μιλήσουμε για λεπτομερή σενάρια. Ε, μία προσεγγιστική εκτίμηση είναι ότι 50 ε, ε, δισεκατομμύρια ευρώ θα διατηρήσουν το σημερινό επίπεδο παροχής ε, δημοσίων αγαθών. Ενώ 10 με 20 δισεκατομμύρια θα μας δώσουν την ευκαιρία για την παροχή περισσότερων δημοσίων αγαθών και σε επίπεδο δασοκομείας κτλ. Νομίζω ότι προς το παρόν πρέπει να κινηθούμε όπως μπορούμε, χωρίς να περιμένουμε ε, για πιο ακριβείς εκτιμήσεις. Ε, με τα 20 δισεκατομμύρια και με συμμετοχή των κυβερνών, νομίζω ότι είναι μια αρκετά καλή εκτίμηση για τις ανάγκες μας. Ε, με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα έχουμε μια ε, βιώσιμη διαχείριση της γης και θα έχουμε τη δυνατότητα να ξοδέψουμε λεφτά και σε άλλες πολιτικές και παράλληλα να μην πέσουν κάτω από ένα επίπεδο οι γεωργοί μας. Αυτά σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Bene, grazie. Valentin Zanert. Ευχαριστώ τον Ολοκληρώσαμε τις παρουσιάσεις των ε, πυρογνών μόνων μας και τώρα ξεκινάμε την ε, συζήτηση. Έχω ένα κατάλογο με όσους ζήτησαν το λόγο. Έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας. Νομίζω ότι θα έχουμε το χρόνο για να δώσουμε το λόγο ξανά ε, και στον Υπουργό Γεωργίας της Σουηδίας για να κάνει κάποιες τελικές παρατηρήσεις. Ξεκινάμε τον κύριο Μόρβεϊ. Κυρία Μόρβεϊ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω ουγγρικά. Νομίζω ότι Καλό θα ήταν η αναθεωρημένη ΠΑΚ να έχει σαφείς προτεραιότητες και ξεκάθαρη φιλοσοφία. Και γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Να δούμε τι προτεραιότητες θα πρέπει να έχει η μελλοντική ΚΑΠ και ποιες αξίες να αντιπροσωπεύει. Έχουμε μια γεωργική πολιτική που φαίνεται ότι επικεντρώνεται στο κέρδος και στα χρήματα. Ε, μοναδικό της μέλημα είναι η ο, προσπόρηση κέρδους. Δεν μας ενδιαφέρει όμως στο μέλλον μια τέτοια ΚΑΠ. Θέλουμε μια ΚΑΠ που να είναι ανθρωποκεντρική και που στόχο θα έχει να εξασφαλίσει μια εξευρεπή επιβίωση στις ε, αγροτικές κοινότητες και να εξασφαλίσει βιωτικές συνθήκες και αξιοπρεπή εισοδήματα στους γεωργούς. Επίσης θέλουμε μια ΚΑΠ που να παραγάγει υγιή τρόφιμα και να σέβεται το περιβάλλον διατηρώντας ε, το τοπίο της υπαίθρου. Η αγροπιστιστική βιομηχανία είναι μία ελίτ μερικές φορές. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές θα πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο και όχι η αγροπιστιστική βιομηχανία. Όπως πολύ προλαλήσατε, θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για τις κλιματικές αλλαγές. Θα πρέπει να ανατρέψουμε, να αντιστρέψουμε αυτή τη διαδικασία ε, επιτάξεις των κλιματικών αλλαγών. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται φορτηγά ή αεροπλάνα για να μεταφερθούν τα τρόφιμα, αλλά αντί να αγοράζουμε τρόφιμα που έρχονται από την άλλη άκρη του κόσμου, γιατί να μην αγοράζουμε τρόφιμα της ντόπια παραγωγής από το διπλανό χωριό, γιατί όσο πιο μακριά ταξιδεύουν τα τρόφιμα, τόσο περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα εκπέμπουν τα μέσα μεταφοράς. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην τόπια παραγωγή και στην παραγωγή που θα βρίσκεται κοντά στην κατανάλωση. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τις κλιματικές αλλαγές και να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου προστατεύοντας το περιβάλλον. Η κατάσταση για τις νέες χώρες είναι πραγματικά ανήθικη και παράνομη. Αυτό ισχύει και για την Ουγγαρία. Είναι πολύ άδικη η κατάσταση για τις νέες χώρες. Η Ουγγαρία υποχρεώθηκε να αναλάβει πολύ ματηρές δεσμεύσεις για την ένταξη, ενώ σε αντάλλαγμα έλαβε πολύ κατακαιρματισμένες ενισχύσεις. Ο Προεδρεύων υπουργό μίλησε για την αδικία που έχει γίνει προς τις νέες χώρες και αυτό με ενθαρρύνει για το μέλλον της ΚΑΠ. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές θα πρέπει να αντιστραφεί αυτή η τάση και να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη μεταξύ παλιών και νέων χωρών. Αλλιώς οι νέες χώρες ε, μέλη θα είναι σαν απικίες των παλιών. Θα χρειαστεί να ξεπουλήσουμε τα εδάφη μας, τα αγροτεμάχια μας, στις πλουσιότερες χώρες που έχουν ε, πολύ πιο υψηλό ΑΕΠ. Αυτή είναι μια κατάφορη αδικία. Πώς σκοπεύετε λοιπόν να διορθώσετε αυτή την αδικία με τα νέα μέτρα της ΚΑΠ. Ευχαριστώ. Καλνιέται. Ε, merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συνθήκη της Λισαβόνα θα τεθεί σε ισχύ και θα επηρεάσει πολύ την, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή μας. Η συζήτηση που ξεκίνησε σήμερα για την κοινή αγροτική πολιτική αποτελεί μόνο, αν θέλετε, την αρχή ενός πολύ δύσκολου δρόμου. Να αναφέρω κάποια αριθμητικά στοιχεία. Οι αγρότες επενδύουν κατά 70% πιο πολύ σήμερα ε, σε σχέση με αυτά που λαμβάνουν από τις ενισχύσεις της ΚΑΠ. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο και γι' αυτό πιστεύω ότι ένας από τους δύο βασικούς στόχους της ΚΑΠΘ είναι να διασφαλίσει μία ισοτιμία, μία δικαιοσύνη μεταξύ των πληρωμών όλων των κρατών μελών. Και αυτό θα πρέπει να γίνει με ισότιμο τρόπο. Θα πρέπει να υπάρχει δίκαιος ανταγωνισμός, προκειμένου οι αγρότες να λειτουργούν υπό ίδιους όρους. Προφανώς ε, όλα τα θέματα που σχετίζονται με δημόσια αγαθά, με την ευημερία των ζώων και το καθεξής θα πρέπει να θεωρηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως και τα πρότυπα προκειμένου να είναι τα ίδια και στις 27 χώρες. Να πω δύο λόγια τώρα για το πώς μπορούν να εντοπιστούν οι δείκτες των ε, άμεσων πληρωμών. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ισχύσουν ιστορικά στοιχεία, ιστορικοί δείκτες. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σημερινή κατάσταση. Θα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους να εντοπίσουμε τα κριτήρια αυτά. Γιατί ούτε καν το κριτήριο των εκταρίων δεν είναι αντικειμενικό για την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας, ωστόσο με τη σωστή αναλογία, προκειμένου όσοι ζουν στην υπαίθρο, όσοι παράγουν α, υγιεινά τρόφιμα και όσοι τα καταναλώνουν, να βρίσκονται σε μια ισορροπία. Δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστό να περιοριστεί η ενίσχυση εις βάρος των ενιαίων πληρωμών μόνο για την Αν παραμείνει το σύστημα του modulation, η χρηματοδότηση που θα προκύψει από τη μείωση των ενιαίων πληρωμών θα πρέπει να κατανεμηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό να γεφυρωθούν τα χάσματα σε επίπεδο παραγωγής προκειμένου να μην βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου κάποιες χώρες θα παράγουν με υψηλά τεχνολογικά μέσα και κάποιες άλλες χώρες, οι καινούργιες ε, χώρες, θα είναι λιγότερο ανταγωνιστικές σε ό,τι αφορά την ε, αγροτική παραγωγή. Γιατί δεν θα έχουν λάβει την ενίσχυση αυτή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να περιορίσουμε λίγο τις παρεμβάσεις για να μιλήσουν όλοι μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. Sí. García. <laughs> Δεν αυτό το έγγραφο που υπάρχει, δεν υπάρχει, μετά πετάχτηκε στα σκουπίδια. Μου θύμισε κάτι που ζήσαμε πριν από μήνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμφανίστηκε ευνίδια ένα έγγραφο, λίγο πριν το διαγνωστικό έλεγχο της ΚΑΠ, που η Επίτροπος μας είπε ότι δεν υπήρχε αλλά μετά δημοσιεύθηκε και ήταν σχεδόν ε, απαράλλακτο το αρχικό έγγραφο που τάχα δεν ήταν ε, επίσημο. Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, σας υπενθυμίζω την πανημία. Σήμερα αναφέρθηκε η σωστή σειρά συζήτησης, ε, αν θα είναι η στόχη πρώτα ή ο προϋπολογισμός. Την τελευταία φορά για τις δημοσιονομικές προοπτικές πρώτα προσδιορίσαμε τους στόχους και μετά τα κονδύλια. Και αυτό μας οδήγησε στη διαφοροποίηση, στη διακύμανση, το modulation. Μπορούμε να έχουμε όλους τους στόχους χιλιετίας για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Αλλά θα συμβεί ότι συνέβη στις Βρυξέλλες το 2005 που έκλεισαν ε, τους κρουνούς της χρηματοδότησης και θα βρεθούμε χωρίς χρήματα για τους φιλόδοξους στόχους. Οπότε από πού θα γίνει οι περικοπές, από την κοινή γεωργική πολιτική. Και έτσι, όπως σας είπα, καταλήξαμε στην διακύμαση, στο modulation. Το θέμα είναι πρώτα να δούμε πόσα διαθέσιμα κονδύλια έχουμε και μετά να το κατανείμουμε στους στόχους. Αλλιώς θα κοροϊδεύουμε και τους πολίτες και τη γεωργία και την κτηνοτροφία, τους γεωργούς και κτηνοτρόφους που περιμένουν τις αποφάσεις μας. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω κυρίως για τον επιστηστικό ανεφοδιασμό. Το θέμα της επάρκειας του διατροφικού ανεφοδιασμού σας φαίνεται σημαντικό, γιατί αντί να παράγουμε θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε μόνο, αν δεν είναι σημαντικό αυτό το θέμα της επάρκειας σε τρόφιμα. Να μην καταλήξουμε να είμαστε εξαρτημένοι από τις τρίτες χώρες για τα σιτηρά μας. Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις του, του ΠΟΕ, ελάχιστα αναφέρθηκαν. Ούτε μίλησε κανένας να ξεπεράσουμε τα κόμπλεξ μας και να επενδύσουμε στην επικοινωνία με τον πολίτη και στην ενημέρωση για το τι εστί και σε τι χρησιμεύει η ΚΑΠ. Γιατί δεν το εξηγεί αυτό η Επιτροπή στους πολίτες. Μόνο εξωτερικές οργανώσεις ε, προσπαθούν να εξηγήσουν τους πολίτες και παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή και ερμηνεία για την κοινή γεωργική πολιτική. Γι' αυτό και πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι η γεωργική πολιτική ουσιαστικά γεμίζει τις τσέπες ορισμένων παραγωγών, κάτι που πόρο απέχει φυσικά από την πραγματικότητα. Συμφωνώ με τον κύριο Μπάκουελ ότι κάποιοι ενισχύσει της θα πρέπει να δίνουν ασφάλεια ε, και όχι αβεβαιότητα στους γεωργούς. Νομίζω ότι οι γεωργοί αξίζουν τις ενίσχυσεις γιατί μας ε, ανεφοδιάζουν με τρόφιμα, εξασφαλίζουν την επιστημιστική ασφάλεια, ε, εξασφαλίζουν την ευημερία των ζώων. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι αμφισβήτο ότι αξίζουν τις ενισχύσεις και δεν θα πρέπει να τις αμφισβητούμε. Άλλωστε οι γεωργοί ε, δεν ε, ε, ανταγωνίζονται σε μια ελεύθερη αγορά και υπόκεινται σε πολύ πιο αυστηρές ρυθμίσεις από αυτές των τρίτων χωρών. Και είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν και σε μια παγκόσμια αγορά. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Όταν εξετάζουμε την ΚΑΠ, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι Ευρωπαϊκή οι Ευρωπαίοι γεωργοί έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Γιατί οι γεωργοί τρίτων χωρών ούτε του ίδιου φόρου πληρώνουν, ούτε τι ίδιε υψηλέ προδιαγραφέ ανιχνευσιμότητα, ευημερία των ζώων ε, κτλ. δεν πληρούν. Αν δεν εξισωθούν οι όροι ανταγωνισμού για όλου του γεωργού, δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από την κοινή γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον ε, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για να ακούσουμε τα τελικά του σχόλια, γιατί θα πρέπει να φύγει αμέσω μετά. Σα Σας ευχαριστώ και που μου δίνετε το λόγο. Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που διοργανώθηκε αυτό το εργαστήριο σήμερα και χαίρομαι που μπορούσα να συμμετέχω. Διαπιστώνω επίσης ε, με ικανοποίηση ότι επικρατεί μεγάλη συνένεση μεταξύ μας. Όλοι θεωρούν ότι το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και είμαι ικανοποιημένος που πολλοί στις ε, συμβολές τους ανέφεραν ότι η Ευρωπαϊκή Γεωργία έχει δυναμικό ανάπτυξης. Είμαι ικανοποιημένος που Μιλάμε για θέσει εργασία στην Ήπεθρο, που υπάρχει ανάγκη για θέσεις εργασία, και επίσης είμαι ικανοποιημένο που πολλοί ομιλητέ ε, στην ε, εισήγησή του ανέφεραν ότι καλό θα ήταν να διοχετευτούν πιο πολλά κονδύλια στα δημόσια αγαθά προκειμένου ο φορολογούμενος με τον τρόπο αυτό να πληρώσει κάτι το οποίο θα τα βρει στο μαγαζιά τελικά. Και νομίζω ότι επίσης ε, με την ε, απλοποίηση, με την απλούστευση θα πρέπει να προκύψει μία πολιτική την οποία θα μπορούμε να εξηγήσουμε στον φορολογούμενο στην Ευρώπη. Θα πρέπει να είναι σαφές, να είναι τόσο σαφές το πρόγραμμα, ώστε τουλάχιστον το καταλαβαίνουν οι αγρότες. Γιατί έχω μιλήσει με πολλούς ε, αγρότες οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν την ε, ΚΑΠ ως ε, έχει σήμερα. Έτσι λοιπόν ε, θα δημιουργήσουμε ευρεία υποστήριξη για την ΚΑΠ και με τους αγρότες, αλλά και σε ό,τι αφορά το ευρύ κοινό, τους φρολογούμενους Και κάτι άλλο. Μην ξεχνάτε τις δυνατότητες που έχουν οι αγρότες στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις ε, ανανεώσιμες ενέργειες. Συμφωνήσαμε στην Ευρώπη σταδιακά να κινηθούμε προς μια κοινωνία απαλλαγμένη από τα ρηκτά καύσιμα. Και εγώ είπα στους ε, αγρότες στη χώρα μου ότι θεωρώ ότι ο δικός σας ο κλάδος θα πρέπει να είναι ο κλάδος ο οποίος πρώτος θα πρέπει να απαλλαχθεί από τα ρηκτά καύσιμα. Επίσης θα ήθελα να θίξω το θέμα των ποσοστώσεων. Σε ορισμένες ε, περιοχές υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν ποσοστώσεις. Αλλά τώρα που ο γαλακτοκομικός κλάδος διανύει κρίση, διαπιστώνω ότι το σύστημα που καθιερώθηκε στον κλάδο αυτό δεν βοήθησε ουσιαστικά τους ε, αγρότες. Δεν είχε αποτέλεσμα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι κάπως αμφιλεγόμενα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις. Αντιθέτως, πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πού φτάνουν τελικά τα χρήματα αυτά. Οι τιμές ε, των τροφίμων για τους καταναλωτές μας ανεβαίνουν, ενώ μειώνονται σημαντικά τα εισοδήματα των γεωργών. Πού καταλήγουν λοιπόν τα χρήματα αυτά. Υπάρχει στρεβλός ανταγωνισμός. Πού βρίσκεται το πρόβλημα στο όλο σύστημα. Και νομίζω ότι και για τους αγρότες, αλλά και για τους φορολογούμενους, για τους καταναλωτές, θα πρέπει να εντοπίσουμε πού ακριβώς διοχετεύονται αυτά τα χρήματα. Και τέλος, θα ήθελα να αναφέρω κάτι το οποίο δεν άκουσα στις εισηγήσεις την κατανάλωση και την ε, παροχή πρωτεϊνών στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το πώς μπορούμε να έχουμε αρκετές πρωτεΐνες. Και πρόκειται για κάτι το απόλυτα επιθυμητό. Νομίζω ότι θα πρέπει να τοποθετηθούμε και σε ό,τι αφορά την ΚΑΠ. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους για την συνάντηση αυτή και ανυπομονώ να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, Εσκύλ. Ε, σε χαιρετίζουμε, αλλά συνεχίζουμε εμείς την συζήτησή μας με τον Στεφάν Λεφόλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τώρα θα μιλήσουμε έτσι μεταξύ μας. Θα είμαι σύντομο γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά και περνάει και η ώρα. Δύο πράγματα θέλω να πω. Πρώτον, πιστεύω ότι θα γίνει μια πραγματική συζήτηση για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο της Γεωργίας. Ο γεωργικός προπολογισμό θα είναι αντικείμενο μεγάλης προσοχής. Ε, κάποιοι θα θέλουν να τον μειώσουν, αλλά ούτως ή θα γίνει μια συζήτηση για τον ίδιο τον κοινωνικό προπολογισμό ε, αναφέρθηκε κατά σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και νομίζω ότι δεν ε, χρήζει λόγος αισιοδοξία. Δεύτερον, άκουσα πολλούς, άκουσα πολλά πράγματα να λέγονται. Πάντως το θέμα που πρέπει να τεθεί είναι πού θέλουμε να πάμε. Όλοι λένε, ε, μιλάμε για τον πριν του στόχου, αλλά τελικά ποιοι είναι οι στόχοι. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, από του στόχου. Αν θέλουμε να έχουμε μια συζήτηση στην ε, Επιτροπή Γεωργία, θα πρέπει να μιλήσουμε για του στόχου καταρχήν. Μιλάμε για το επιστηστικό θέμα. Η Επίτροπος το είπε, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι πεινάνε στον πλανήτη. Θα έλεγα 18 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πεινάνε επίσης, μην ξεχνάμε και αυτούς. 18 εκατομμύρια λιμοκτώνουν επίσης. Επομένως το θέμα της διατροφής είναι στην, ε, στον πυρήνα της συζήτησης, ναι. Ε, το περιβαλλοντικό θέμα, όλοι μιλούν γι' αυτό. Μιλάμε ε, Επινοούμε και ένα τρίτο πυλώνα για το, τα περιβαλλοντικά θέματα. Με αυτόν τον τρόπο όμω θα επιληθεί το πρόβλημα. Αν είναι ένα μείζον θέμα ε, για το μέλλον, όχι μόνο τη Ευρώπη, αλλά και του πλανήτη, θα πρέπει να έχουμε τα μέσα για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Το οικονομικό και κοινωνικό θέμα. Όλοι μιλάνε για την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα. Εγώ θέλω να είναι ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Γεωργία, αλλά δεν θέλω να έχουμε μόνο αυτό το κριτήριο. Ε, μόνο με αυτόν τον τρόπο να κρίνουμε τις επιδόσεις της γεωργίας. Υπάρχει το κοινωνικό στοιχείο, η απασχόληση που εξασφαλίζει η γεωργία και το θέμα της ε, ποικιλομορφίας της γεωργίας, της ε, γαλλικής, ε, παύλα ευρωπαϊκής γεωργίας, τσαμπών, τυρί, σε όλη την Ευρώπη, όλα αυτά. είναι γνωστά. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε στόχους, θα πρέπει να είμαστε οικονομικά ανταγωνιστικοί, οικολογικά πάρα πολύ καλή και, και κοινωνικά επίσης ε, να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να είναι σε θέση να θρέψει τον κόσμο, θα πρέπει να απαντήσει στο περιβαλλοντικό πρόβλημα και θα πρέπει να απαντήσει και στο ερώτημα του τι Ευρώπη θέλουμε, τι εικόνα της ευρωπαϊκής ε, γης, του ευρωπαϊκού τοπίου θέλουμε να προβάλλουμε. Αυτό είναι το θέμα. Και να πω και κάτι πιο τεχνικό. Αυτό σημαίνει ότι αντί να μιλάμε για πρώτο και δεύτερο πυλώνα, ε, για το, την πασαρέλα μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα, πώς θα ρυθμίσω το α και το β, ε, θέλουμε, πρέπει να πούμε, θέλουμε πολιτική για την Ήπεθρο. Όχι, θέλουμε πολιτική γεωργική, επισητιστική και, για και πολιτική για την Ήπεθρο. Και όλες οι γεωργικές ενισχύσεις θα πρέπει να έχουν αυτούς τους στόχους. Εγώ είμαι υπέρ αυτό που είπε ο κ. Σατελιέ και υπέρ αυτών που είπε ο πρώτος ομιλητής. Θα πρέπει η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική να εξασφαλίσει το πέρασμα της Ευρω... μιας γεωργίας όπως την ξέρουμε μέχρι στιγμής προς μια γεωργία που ε, εξασφαλίζει και τη γεωργική διάσταση και την επιστηστική διάσταση και την περιβαλλοντική διάσταση. Αν λοιπόν θέλουμε να, έχουμε, να υλοποιήσουμε κάποιους στόχους, θα πρέπει να έχουμε και τα μέσα. Θέλω να υπάρχει ένας μεγάλος πυλώνας λοιπόν, ε, γεωργικός, περιβαλλοντικός και κοινωνικός, που θα μας εξασφαλίσει το πέρασμα ε, προς τη γεωργία που θέλουμε αύριο. Ευχαριστώ Στεφάν για την έμπλεη πάθος παρέμβασή σου. Προφανώς ε, συμφωνούμε μεταξύ μας, το λέμε εδώ μεταξύ μας βέβαια. Αλλά εμεί είμαστε άνθρωποι που θα έχουμε τελικά και ευθύνε για αυτά τα θέματα. Οπότε αυτό που λέμε έχει νόημα. Το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής απαιτεί συνέχεια αλλά και αλλαγές. Αλλαγές ως προς την εφαρμογή του γεωργικού Συμβολίου, Συμβολέου συγγνώμη, και τη λήψη υπόψη των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης και του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να είναι και δίκαιη η κοινή γεωργική πολιτική και να δούμε πώς αξιοποιείς τα διάφορα κονδύλια. Ο προϋπολογισμός της ε, ε, ΚΑΠ είναι 30% ε, της, του κοινωτικού προϋπολογισμού, αλλά μόνο 0,3% του ΑΕΠ της Ένωσης. Ενώ είναι κοινωτική πολιτική, χρηματοδοτείται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά κυρίως χρηματοδοτείται από τα κράτη-μέλη. Και εκεί έγκυται το πρόβλημα. Αυτό το ποσοστό τι θα γίνει, πώς θα αλλάξει μετά το 2013. Θα μειωθεί, η ανάγκη των αλλαγών είναι εμφανής. Αλλά τα γεωργικά εισοδήματα σε, όλα τα, όλη την Ένωση είναι χαμηλότερα από τα εισοδήματα άλλων παραγωγικών κλάδων και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η εμπειρία μας έδειξε την εξάρτησή μας στην περίπτωση της ενεργειακής κρίσης από τις εισαγωγές του αερίου, του φυσικού αερίου. Έχουμε και τη χρηματοπιστωτική κρίση. Δεν θέλουμε αντίστοιχη εξάρτηση για τα τρόφιμα. Άλλωστε διαπιστώσαμε ότι μόνη της χρηματοπιστωτική αγορά δεν μπορεί να αυτορυθμιστεί. Και μην ξεχνάτε ότι οι γεωργοί εξαγαρτώνται από τη βιολογία, από τις κλιματικές αλλαγές. Δεν υπάρχουν σταθερές συνθήκες για την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. Οπότε και μόνο ο προσανατολισμός της αγοράς δεν εξασφαλίζει τη σταθερότητα στην κοινοτική αγορά. Επίσης, το κόστος των κλιματικών αλλαγών. Το κόστος της χρηματοπιστωτικής κρίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Γιατί τα ποσά που θα αφιερωθούν στη Γεωργία δεν λαμβάνουν υπόψη όλες αυτές τις κρίσεις. Πώς θα αντιμετωπίσουν οι Γεωργοί μόνοι τους όλα αυτά τα δεινά. Και το, η γεωργία απορροφά τόσα κονδύλια όσο και αυτά που προσφέρει, από αποδίδει. Υπάρχει το θέμα της διαχείρισης του ύδατος. Η γεωργία θα πρέπει να συμβάλλει στην εξορθολογισμό της διαχείρισης του ύδατος. Επίσης, τι θέλουμε να στηρίξουμε, τα εισοδήματα, την ανταγωνιστικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, να προστατεύσουμε τα εισοδήματα των γεωργών, την ασφάλεια του επιστηστικού εφοδιασμού. Αναφέρθηκε η στοχευμένη στήριξη. Ναι, αλλά πώς θα την, επιδι... πώς θα την υλοποιήσουμε και πώς θα την ελέγξουμε. Πώς θα τη χρηματοδοτήσουμε ή πώς θα ε, αξιολογήσουμε το δημόσιο αγαθό που προκύπτει από τη Γεωργία. Έχω πολλά θέματα που με απασχολούν, αλλά θέλω να, να περιοριστώ σε δύο. ΠΟΕ, θα πρέπει να κινητοποιήσουμε την παγκόσμια πολιτική για τη γεωργία. Γιατί παγκόσμια χώρα απαιτεί και παγκόσμια προσέγγιση για τα γεωργικά ζητήματα. Επίσης, πολιτική συνοχής και ΚΑΠ. Η πολιτική της υπαίθρου. Μερικές φορές τα κονδύλια που αφαιρώνται στη γεωργία εξυπηρετούν άλλους στόχους συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε μια κοινή και ισχυρή γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπε και η Επίτροπος. Και μην κοφεύετε στη φωνή των νέων χωρών που έχουν ε, ε ιδιαιτερότητες στη γεωργία τους. Μερικές φορές ε, η Κομισιόν έκανε το κεφαλιού της και δυστυχώς δεν είχαμε πάντα θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Κύριε Μαγκίνες. Έχουμε άλλα 7-8 άτομα. Θα ήθελα να επιταχύνουμε τώρα σε αυτή την τελική ευθεία. Η ε, κύριε Μαγκίνες. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Ε, αν και ελπίζω να το ξαναθίξουμε το θέμα αυτό. Καταρχάς, ε, είναι κρίσιμο το θέμα αυτό. Κατά δεύτερον, πιστεύω ότι η διαρροή, αν θέλετε, του εγγράφου αυτού των επίσημου έγινε υπό τον όρο ότι η κοινότητα και εμείς ως πολιτικοί θα το λάβουμε προκειμένου όταν θα δημοσιευτεί επίσημα να φανεί λιγότερο ακραίο. Να αντιδράσουμε λιγότερο θυμωμένα, αν θέλετε. Γιατί έτσι γίνεται συχνά. Διαρρέει κάτι χειρότερο για να ικανοποιηθούμε με το καλύτερο. Κατά δεύτερον, ήταν κάπως ακαδημαϊκές οι συζητήσεις, οι παρουσιάσεις, αλλά πολύ χρήσιμες. Δεν αποδέχομαι τις επικρίσεις αναφορικά με την ΚΑΠ που ακούστηκαν εδώ στην αίθουσα αυτή και που φαίνεται να αποδέχεται σαν Ευαγγέλιο η Επιτροπή μας. Και νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε με σαφήνεια ότι το κοινό δεν είναι τόσο κριτικό πια για την ΚΑΠ όσο υπονοείται στον τύπο και να προσέξουμε, μην αναπτύξουμε μία πολιτική βάσει της τελευταίας έκθεσης στον τύπο για τις πληρωμές ε, στα πλαίσια της ΚΑΠ βάσει βάση της τελευταίας τηλεοπτικής εκπομπής. Ήμουν δημοσιογράφος και είμαι πολιτικός τώρα και καταλαβαίνω και τις δύο πλευρές. Είναι πολύ επικίνδυνο αν η πολιτική μας ε, ακολουθήσει την τελευταία αναταραχή, αν θέλετε, στον τύπο. Νομίζω ότι το κοινό κατανοεί τα θέματα της ε, γεωργικής πολιτικής και την υποστηρίζει και κατανοεί και ότι τις αποτυχίες της αγοράς. Ένας από τους ε, προλαλήσαντες ανέφερε το εξής, ότι η κοινωνία εκτιμά ιδιαίτερα τις υπηρεσίες, αλλά να πω ότι δεν ε, Τιμολογία, αν θέλετε, απαραίτητα τις υπηρεσίες αυτές η κοινωνία. Αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς ως πολιτικοί και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στις ε, συζητήσεις αυτές για την ε, επισητιστική ασφάλεια. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική και ήμουν υπεύθυνη για την σχετική έκθεση στην τελευταία θητεία. Η ενιαία πληρωμή στα αγροκτήματα είναι ένας άμεσος τρόπος για την παροχή χρημάτων στους ε, αγρότες και να κάνω μια ερώτηση και ένα σχόλιο. Όσοι από προχωρήσουν σε, πλήρα, σε πλήρη αποδέσμευση, δεν θα πρέπει να τιμωρηθούν για την αποδέσμευση αυτή. Να σκεφτούμε λοιπόν μήπως μπορούμε να ανανεώσουμε την περίοδο αναφοράς. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή ως περίοδο αναφοράς μια πιο πρόσφατη περίοδο. Αυτό συζητιέται επί τόπου. Θα θέλετε να σχολιάσετε για το θέμα αυτό. Θα περιοριστώ σε αυτά, Πρόεδρε, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι ομιλητές και θα το ξανασυζητήσουμε άλλωστε και στο μέλλον το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Γκαρσία Τώρα σε τόσο προχωρημένο στάδιο της συζήτησης δεν υπάρχει τίποτα καινούριο πια. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση για το εργαστήριο μελέτης. Και φυσικά ακούσαμε πολλές σκέψεις. Θα μπορούσαμε να τις αναλύσουμε και έχουν πολλές χρειές καθεμία. Η Επίτροπος, για παράδειγμα, ξεκίνησε πολύ ευφυώς με δύο διαπιστώσεις. Είπε ότι θα πρέπει να ταχθούμε υπέρ μιας ισχυρής ε, και κοινή γεωργικής πολιτικής, η οποία όμως θα πρέπει να τροποποιηθεί. Και λέω το είπε έξυπνα, γιατί ως προς αυτό συμφωνούμε. Η δυσκολία όμως ε, θα προκύψει αργότερα, όταν θα κρυθούμε να αποφασίσουμε για το ποιε αλλαγέ θα θεσπίσουμε στην κοινή γεωργική πολιτική. Αναφέρθηκε η προστιθέμενη αξία της γεωργίας και σε άλλους τομείς, όπως του περιβάλλοντος, στη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, ε, στην σταθεροποίηση του πληθυσμού στις αγροτικές ζώνες και στη μη εγκατάλειψη των ζώνων αυτών. Όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη για να αποφασίσουμε για το ποιες αλλαγές θα προτείνουμε στην ΚΑΠ. Έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις τώρα. Σε ό,τι αφορά την ενιαία ενίσχυση. Αναφέρθηκε πολλές φορές το θέμα αυτό. Το επισήμανε και ο Προεδρεύων. Μίλησε για τις αρνητικές συνέπειες της άμεσης ενίσχυσης και εμπειρογνώμονε το ανέφεραν, προβλήματα που απορρέουν από την ενιαία ενίσχυση. Το θέμα είναι τι αλλαγέ θα γίνουν στο σύστημα αυτό. Δεν θα πρέπει όμω να μιλούμε μόνο για τα μειονεκτήματα αυτού του καθεστώτο ενιαία ενίσχυση, αλλά να δούμε ποια ήταν και τα πλεονεκτήματά του. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι πολλοί παραγωγοί, γεωργοί και κτηνοτρόφοι τη Ένωσης κατάφεραν χάρη σε αυτό το καθεστώ ενιαίας ενίσχυση να επιβιώσουν και να διατηρήσουν την, την ε, γεωρική τους δραστηριότητα. Μα το είπαν ότι χάρη στην ενιαία αυτή ενίσχυση μπορώ να διατηρήσω την ε, εκμετάλλευσή μου. Αλλιώ θα είχα κατεβάσει τα ρολά και θα μετακόμιζα σε μια πόλη. Ας ε, βάλουμε λοιπόν στην πλάστιγκα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης για να δούμε τι αλλαγές χρειάζονται, αλλά να μην εστιαζόμαστε μόνο στα αρνητικά και να αμελούμε τα θετικά. Πολλές φορές αναφέρθηκε στην απογευματινή συζήτηση η ανάγκη ο Ευρωπαίος πολίτης να κατανοήσει, να αντιληφθεί και μιλήσαμε για τον Ευρωπαίο πολίτη πώς φορολογούμενος θα πρέπει να καταλαβαίνει πώς αξιοποιούνται τα φορολογικά του, φορολογική του φορά. Θα πρέπει επίσης να εξηγήσουμε στον Ευρωπαίο πολίτη τι κάνουμε με τον κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά και τι κάνουμε με τα κονδύλια και γιατί πληρώνει για ένα λίτρο γάλακτος και ένα κιλό κρέατος τα διπλάσια από ό,τι πλήρωνε πριν από μερικά χρόνια, ενώ η ενίσχυση που λαμβάνει ο Γιώργος έχει μείνει αμετάβλητη. Όλα αυτά θα πρέπει να τα εξηγήσουμε. Η, συζήτηση είναι περίπλοκη, έχει πολλές διαστάσεις. Θα πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε την ευθύνη που μας βαρύνει αυτή τη στιγμή και παίζουμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και ελπίζω ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε σαφείς απόψεις και τα έγγραφα όπως το περίφημο έγγραφο που διέρευσε και κατέληξε στα σκουπίδια είναι βάσεις για συζήτηση που θα πρέπει να μας αφυπνίζουν για την πραγματικότητα γιατί θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη μας τη στιγμή που καθορίζουμε το μέλλον χιλιάδων γεωργών και κτηνοτρόφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ που πήρατε αυτή την πρωτοβουλία των εργαστηρίων αυτών για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για ένα θέμα το οποίο θα είναι πολύ σοβαρό. Ε, θα ήθελα να παραμείνω σε επίπεδο αρχών και να ε, κρατήσω δύο-τρεις ιδέες από όλα όσα ακούστηκαν σήμερα. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι δεν πιστεύω ότι είμαστε αποτελεσματικοί απέναντι στην κοινή γνώμη όταν λέμε ότι α, μπορούμε με μία μόνο πολιτική να υλοποιήσουμε διάφορους στόχους. Θα πρέπει να χτίσουμε μια πολιτική κοινή επισητιστικής ασφάλειας. Αν ε, πούμε στον πολίτη ότι ο στόχος μας είναι ε, να υποστηρίξουμε τους γεωργούς, τον, τον οποίον αριθμός μειώνεται, ε, στην πραγματικότητα είναι σαν να υποστηρίζουμε μόνο μια κατηγορία. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η γεωργία με την ασφάλεια που μας δίνει, με την ανεχνησιμότητα των, των τροφίμων, ε, διαχείρισης του, ε, του τοπίου, ε, του περιβάλλοντος κτλ. Νομίζω ότι ε, φυσικά, ο τρόπος που παράγουμε τα τρόφιμά μας σχετίζεται με το περιβάλλον. Το θέμα του περιβάλλοντος είναι πολύ ευρύτερο από το θέμα της γεωργίας. Θα πρέπει να διαχωρίσουμε αυτές τις πολιτικές. Δεύτερον, είπαμε πάρα πολλά για τον πρώτο πυλώνα, τον δεύτερο πυλώνα. Άκουσα το πώς εξηγήσε ο Στεφάν Λεφών, ότι πέρα από αυτά θα πρέπει να διαρωτηθούμε για τους στόχους της ΚΑΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με αυτά που είπαν πολλοί ομιλητές, ομιλητές κυρίως με τον κ. Σατελία, που είπε να μία από τις ελάχιστες πολιτικές που είναι πραγματικά ευρωπαϊκές, διατρήσουμε ως τέτοια. Και ας αρχίσουμε να τη συγκρίνουμε μαζί με άλλες με άλλε πολιτικέ που δεν είναι μόνο ευρωπαϊκέ. Όταν ακούω να λέτε ότι κοστίζει ακριβά η ευρωπαϊκή γεωργία, η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική, να μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχουν, ε, ε, δεν υπάρχουν εθνικοί προπολογισμοί για διάφορε πολιτικέ. Ενώ εδώ πέρα πραγματικά έχουμε συνεισφέρει όλοι στον ίδιο κορβανά. Ε, θέλω να θέσω δύο ερωτήματα. Καταρχά, ε, ένα τμήμα των κανόνων που υπάρχουν για να υποστρίξουμε τον, το περιβάλλον και τον καταναλωτή. Ε, Εν συνεχεία, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν το κάναμε για να πιέσουμε τους γεωργούς και για να προστατεύσουμε τον καταναλωτή. Οι κανόνες για την προστασία του καταναλωτή ε, θα πρέπει να ε, χρησιμεύουν ως εμπόδιο για ξένα προϊόντα τα οποία θέλουν να μπουν στην αγορά μας ε, με, την, με τον ισχυρισμό ότι σέβονται τους δικούς μας κανόνες. Αν εξηγούμε στον γεωργό από την Ιταλία ε, ή τη Γαλλία, ας πούμε, ότι πρέπει να κάνει αυτά τα πράγματα με αυτούς τους κανόνες, ε, γιατί να μπαίνουν προϊόντα από τον ε, Βραζιλιάνο, ας πούμε, παραγωγό που δεν σέβεται αυτού τους κανόνες. Ε, το θέμα είναι τι κάνουμε. Θα πρέπει να διαρωτηθούμε ε, και δεν θα πρέπει να μπούμε σε ένα παιχνίδι, σας δίνουμε τόσα και εσείς ξοδεύετε τόσα. Θέλω να τελειώσω με το εξή. Γιατί ήδη είπα πολλά δεδομένε τη ώρα. Αφορά τι διαπραγματεύσει των ΠΟΕ. Ε, εδώ και πολλές συνεδριάσεις, ακούμε διάφορες εκθέσεις, ακούσαμε στην, το Σεπτέμβριο ε, μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση για, για μια έκθεση που ακούστηκε στην, στο γύρο της Ντόχα για την παραγωγή του κρέατος θα πρέπει να ψάξουμε δε και καλά να συμφωνήσουμε σε επίπεδο ΠΟΕ, εάν το ερώτημα είναι απλώς πώς θα περιορίσουμε τις αρνητικές συνέπειες. Δεν μπορούμε από τη μία να λέμε ότι ο φιλελεύθερισμός δεν είναι μια λύση για τα πάντα και από την άλλη να μην θέσουμε το ερώτημα μήπως το συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να ξαναδούμε με ποιον τρόπο μπήκαμε σε κάποιες διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ τον κύριο Μπεσού, ο Ζωζέ Μπουβέ και εν συνεχεία άλλες τρεις παρεμβάσεις και κλείσαμε. Μπερδέστηκα με τα κουμπιά μια στιγμή. Με μεγάλη χαρά ακούω τον συνάδελφο τον κύριο Μπεσού που κάνει αυτή την παρέμβαση. Ε, φαντάζομαι, ε, αν είχαμε γνωστεί νωρίτερα, το 1900 99 ε, θα μπορούσαμε να είμαστε μαζί στο Σιάτλ. Ε, θα είχαμε κερδίσει χρόνο. Ε, δεν πειράζει, ίσως όμως θα βρεθούμε στη Γενέβη στο τέλος του μήνα. Αν υπάρχει νομιμότητα σήμερα για την ΚΑΠ, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Υπάρχει νομιμότητα. Η ΚΑΠ όπως λειτουργεί σήμερα δεν νομίζω ότι έχει νομιμότητα. Σε ό,τι αφορά την κατανομή των ενισχύσεων κοινωνικά δεν είναι δίκαιη. 80% ε, των γεωργών ε, αποκλείονται, οικολογικά είναι καταστροφική γιατί δεν έχει ε, σταματήσει την εκβιομηχάνηση της γεωργίας. Βλέπουμε πώς μολύνονται τα νερά μας και οι γης μας και οικονομικά είναι παράλογοι γιατί σήμερα είμαστε σε μια παράδοξη κατάσταση όπου οι τιμές των γεωργικών προϊόντων είναι αποσυνδεδεμένες από την οικονομική πραγματικότητα της παραγωγής. Σήμερα δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ένας γεωργός στην Ευρώπη, ο οποίος είναι ικανός να παράγει με την τιμή της παγκόσμιας αγοράς. Μας επιβάλλεται μια τιμή απλώς. Δεν υπάρχει ε, κανένας γεωργός που μπορεί να παράγει με την τιμή αυτή της παγκόσμιας αγοράς. Όντως λοιπόν υπάρχει ανάγκη να νομιμοποιήσουμε την ΠΑΚ. Γι' αυτό να, την ΚΑΠ. Γι' αυτό να ξανα δούμε τα θεμελιά της. Τα θεμελιά, τα είπαμε, ε, το δικαίωμα να τραφούμε, να παράγουμε την τροφή μας, τα τρόφιμά μας, ε, ίδια πραγματικότητα για τις υπόλοιπες χώρες, ε, ποιότητα παραγωγής, βιοπικιλότητα, κλίμα, απασχόληση. Η απασχόληση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Στη βιολογική γεωργία ε, για την ίδια έκταση είναι επί 30% περισσότερε θέσει απασχόληση. Ξέρουμε ότι οι τρόποι παραγωγή μπορούν να προσανατολίσουν τι θέσει απασχόληση προ συγκεκριμένου τομεί. Πρέπει να το ε, έχουμε υπόψη μα αυτό. Μην ξεχνάμε την ε, λογική που, με την οποία ξεκινήσαμε το 1992. δημιουργήσαμε μια ΚΑΠ που ο στόχος της ήταν να ικανοποιήσουμε εκείνους που μπαίνουν στο παιχνίδι της βιομηχανικής παραγωγής. Ε, μιλάμε για το 7-8% ε, τα, τα της, ε, των εμπορικών ανταλλαγών. Αυτό δεν έχει νόημα σήμερα. Θα πρέπει να βρούμε νέα εργαλεία. Και νομίζω ότι θα αποκτήσουμε νομιμότητα στη γεωργική πολιτική εάν ε, έχουμε στόχους οι οποίοι είναι τριών ειδών. Θα πρέπει να φύγουμε από αυτή την αποσύνδεση ε, της παραγωγής και της ε, στήριξης. Αυτό πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση από τη συνένεση που υπήρχε πριν από λίγα χρόνια. Αλλά αυτή η αποσύνδεση δεν έχει σαν αποτέλεσμα να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, αλλά να κρύψουμε τις επιδοτήσεις από το πορτοκαλί κουτί στο πράσινο κουτί. Αλλά πολιτικά δεν είναι αποτελεσματικό αυτό. Θα πρέπει να ξαναδούμε λοιπόν ε, πώς θα ελέγξουμε την παραγωγή και να μην διαλύσουμε αυτά τα εργαλεία. Παραδείγματο χάρη οι γαλακτοκομικέ ποσοστώσει, αλλά υπάρχουν και, άλλες, και άλλα τέτοια εργαλεία. Θα πρέπει να καθορίσουμε τι τιμέ. Ε, το είπαμε για τα γαλακτοκομικά, αλλά το να καθορίσουμε τιμέ ε, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο δυνάμει του κόστου παραγωγή ε, στι περιοχέ, τις πιο ευνοϊκές αγρο κλιματικά και οι βοήθειε να δίνονται ανάλογα με τα φυσικά μειονεκτήματα. Αυτή η πολιτική ποτέ δεν εφαρμόστηκε και μπορεί να προωθηθεί. Μπορεί να είναι ένα στόχο τη ΚΑΠ. Και τέλο, για να μην μακρηγορήσω, θα πρέπει να υποστηρίξουμε τρόπου παραγωγή που είναι ε, οικολογικά υπεύθυνοι και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε για να αποβιομηχανοποιήσουμε κάποιες παραγωγές. Γιατί δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε μια βιομηχανική γεωργία η οποία για να υπάρξει ε, εισάγει 20 ε, εκατομμύρια ε, τόνους από την Λατινική Αμερική. Ε, οικονομικά και πολιτικά ε, δεν έχει νόημα. Αν θέλουμε να, να καλύψουμε τις ανάγκες των καταναλωτών, των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και καταρχήν των γεωργών, θα πρέπει να αλλάξουμε την γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ, Ζωζέ. Και άλλες δύο παρεμβάσεις. Πίτερ και ο Herbert. Ο ευχαριστώ Πρόεδρε. Τέσσερι σύντομε παρατηρήσει καταρχά ε, για τον επίσημο έγγραφο, το οποίο θα εξαφανιστεί στον, κλάδο, στον κάβο των ε, απορριμμάτων. Φιλικά, πειρά. Ε, θα πρέπει πάντα να εξετάζουμε και με τα δύο μάτια τα θέματα προϋπολογισμού. Και υπάρχουν ε, κάποιες ομάδες που απλά θέλουν να αφαιρεθούν τη χρηματοδότηση. Αυτό βγάζω εγώ συμπέρασμα. Κατά δεύτερα, για την κοινή αγροτική πολιτική. Πιστεύω ότι η κοινή αγροτική μας πολιτική δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο που να έχει εξαντλήσει το δυναμικό της. Κάποιος συνάδελφος το είπε στην αρχή της συζήτηση ότι μιλάμε για 500 εκατομμύρια άτομα για υγιεινά τρόφιμα, σωστή γεωργία και αυτό που ξεχνάνε πολύ είναι ότι είναι υγιείς οι αναλογίες κατά τρίτον για τις ε, αποσυνδεδεμένες πρημοδοτήσεις. Με ενοχλεί το γεγονός ότι μιλάμε πάντα για πίεση του κοινού, ότι οι αγρότες παίρνουν χρήματα και δεν κάνουν τίποτα. Όχι, υπάρχει πολλαπλή συμμόρφωση. Και δεν έχουμε καταρθώσει να εξηγήσουμε στο κοινό ότι οι αγρότες πρέπει να δίνει και ένα αντάλλαγμα για την πρημοδότηση αυτή. Έγινε η αποσύνδεση από το προϊόν, γιατί παλιά παρήγαν πολύ μόνο το συγκεκριμένο προϊόν που ε, έφερνε χρήματα και τώρα πλέον έχουμε θέσει όρους συγκεκριμένους. Αν μας λένε οι έρευνες ότι θα αρκούσαν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυτό λένε και οι σχετικοί μελέτες. Και κατά τέταρτον να πω ότι η δεύτερος πυλώνας, ο περίφημος δεύτερος πυλώνας, έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα, το οποίο συνδέεται με τη συγχρηματοδότηση. Και οποιοδήποτε το προβάλλει ως πανάκια το μέσο αυτό, δεν θα πρέπει να ξεχνάει την συγχρηματοδότηση, η οποία εξαρτάται από το αν έχουν πόρους και οι χώρες. Να το προσέξουμε λοιπόν αυτό. Μην ε, καταλήξουμε σε μια καινούρια άδικη, αθέμητη κατάσταση. Να χρησιμοποιούν δηλαδή τις ενισχύσεις αυτές μόνο τα κράτη που μπορούν. Ευχαριστώ, ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που έγινε σήμερα αυτή η συζήτηση και νομίζω ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας, όλης, μιας μεγάλης διαδικασίας και θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο χρειαζόμαστε μια εκβάθρον μεταρρύθμιση. Θυμάμαι ότι πριν από μια δεκαετία κάναμε τρεις μεγάλες ε, ε, αναθεωρήσεις, μεταρρυθμίσεις. Και θέλουμε τώρα να συνεχίσουμε. Να αναρωτηθούμε όμως